to start because at we will have the ε, Διότι περιμένουμε την Βελγική Προεδρία που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ε, ημερήσια διάταξη. Ε, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει καμιά αντίρρηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν κάποιες εβδομάδες ορίστηκα η Συγήτρια και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε μία συμφωνία σχετικά με την ε, βιομηχανική πρόοδο. Η πρότασή μου όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ήταν να γίνει μία πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων ε, για την ΆΚΑ πριν τις διακοπές, δηλαδή τούτη τη βδομάδα. Το θέμα αυτό όμως δεν βρίσκεται στην ημερησία διάταξη, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Καταλαβαίνω ότι με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και πολλές αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε. Ε, σέβομαι την απόφαση των συντονιστών μας. Ωστόσο προτείνω, κύριε Πρόεδρε, και στου συντονιστές μας το θέμα αυτό να μπει στην ημερήσια διάταξη μετά τις διακοπές, λέει το Σεπτέμβριο. Πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων χωρί καθυστέρηση, λαμβάνοντα ιδιαίτερα υπόψη τι ε, πρόσφατε εξελίξει, τι δηλώσει χθε ε, τη Βαρόνη Άστον. όσον αφορά ε, το εμπόριο ανθρώπων, τη θέση του Ισραήλ καθότι είναι καθαρά τεχνική η συμφωνία αυτή και επειδή είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην καθυστερήσει την διαδικασία όσον αφορά τα ε, φάρμακα. Τονίζω και πάλι, το θέμα δεν είναι τα όπλα, είναι τα φάρμακα. Μιλάμε για ζωές ανθρώπων. Σας παρακαλώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε να στηρίξετε το αίτημά μου και την πρότασή μου να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ΆΚΑ τον Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας στο θέμα που αναφέρατε. Ε, με ομόφωνη απόφαση των συντονιστών συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή της πολιτικής σας ομάδας και με την έγκρισή μου ε, δεν θα αλλάξω την απόφαση αυτή, εκτός εάν όλοι οι συντονιστές ε, συμφωνήσουν κάτι αντίθετο, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του συντονιστή της πολιτικής σας ομάδας. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις, εγκρίνεται η ημερησία διάταξη, καθότι ο καθότι η συνάδελφός μας ε, ε, αντιπρόεδρος δεν βρίσκεται εδώ μαζί μας και μου είπε ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα. Το θέμα υπαριθμών 3 της ημερήσιας διάταξης, ένδειξη της χώρας καταγωγής, θα συζητηθεί αύριο μετά τη ψηφοφορία. Αντί για το σημείο 3, θα συζητήσουμε το ε, θέμα υπαριθμών 3, γνωμοδότηση για τις ε, πτυχές αστικού εμπορικού ε, οικογενειακού και ε, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράση για την εφαρμογή του προγράμματος Στοκχόλμης, για το οποίο η εισηγητής είναι ο συνάδελφος Τζο Higgins από την ΚΟΕ. Να πάμε στο θέμα 2 της ημερησίας διάταξης, ανακοινώσεις του Προέδρου. Ε, όπως γίνεται συχνά, θα ε, μεταδοθεί η ε, συνεδρίασή μας ε, στο διαδίκτυο. Βλέπετε στους φακέλους σας κάποια θέματα. Όποιος ενδιαφέρεται για κάποιο συγκεκριμένο θέμα μπορεί να απευθυνθεί στην γραμματεία. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι για το 2011 όλες οι επιτροπές συμπεριλαμβανομένες της δικής μας θα πρέπει να συμπεριλάβουν συνεδριάσεις Δευτέρες και Πέμπτες ε, στο ημερολόγιο τους. Η γραμματεία Ίντα προτείνει να αυξήσουμε τον ε, αριθμό ε, των τριών συνεδριάσεων μισής ημέρας στα δύο τρίτα ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον κανόνα αυτόν με τη θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, η σχετική πρόταση θα υποβληθεί ε, στην επόμενη συνεδρίασή μας και θα δούμε τότε και πρόταση της Γραμματείας. Άλλο θέμα που, για το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω είναι το αίτημα της ΙΜΚΟ της Επιτροπής Εσωτερικού Εμπορίου για γνωμοδότηση. Ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής αυτής, της ΙΜΚΟ, μου έστειλε επιστολή ζητώντας μας ε, να ε, αναβάλουμε το ημερολόγιο για την πρόταση κανονισμού για την χώρα καταγωγής ώστε να μπορέσει η ΙΜΚΟ να συντάξει γνωμοδότηση. Μίλησα με την εισηγήτρια, την ε, κυρία Μουσκαρδίνη και όλους τους τους συντονιστές και όλοι συμφώνησαν να απαντήσουμε αρνητικά και αυτό έκανα άλλωστε λόγω του ότι το θέμα αυτό το οποίο έχει κολλήσει από το 2005 Ε, θέλουμε να ε, περάσει ε, επί Βελγικής Προεδρίας. Η Επιτροπή μας θα ήθελε να φροντίσει η συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση να επιτευχθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα πριν το τέλος δηλαδή της Βελγικής Προεδρίας. διαβεβαίωσα τον συνάδελφό μας, τον κύριο Μάρκον Χάρπορ, πρόεδρο της ΙΜΚΟ, ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του στο μέλλον και τον καθησύχασα λέγοντάς του ότι η ΙΜΚΟ ήδη είχε την ευκαιρία να ε, εκφραστεί για το θέμα αυτό στο νομοθετικό ψήφισμα που έχει να κάνει με ε, τα ονόματα υφασμάτων ε, και τις προδιαγραφές για προϊόντα υφασμάτων. Όπως συμφωνήσαμε, προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 11, το οποίο αντικαθιστά το 3. Το σημείο 11 έχει να κάνει με τις ε, πτυχές εμπορικού δικαίου του σχεδίου δράσης ε, για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοχόλμης ε, για την ελευθερία ασφάλεια και δικαιοσύνη. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Τζούρι ετοιμάζει έκθεση πρωτοβουλίας για διάφορες πτυχές δικαίου του σχεδίου δράση για την εφαρμογή του προγράμματος Στοκχόλμης που εκδόθηκε στις 20 Απριλίου φέτος. Το σχέδιο δράσης στόχο έχει τη δημιουργία μιας περιοχής ελευθερία ασφάλεια και δικαιοσύνη για τους πολίτες Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή Τζούρι είχε κάποιε ερωτήσει σχετικά με την ε, προσέγγιση και εναρμόνιση των ε, νομοθεσιών, την ε, τυποποίηση κάποιων νομικών ενιών και την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων. Τα θέματα αυτά συνδέονται με διάφορα θέματα που συζητάει η ίντα, μεταξύ άλλων τα πλαστά προϊόντα, τα διανοητικά δικαιώματα, το παράνομο εμπόριο όπλων, ε, θέματα σύγκρουσης δικαίου κλπ. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το συνάδελφο στον συνάδελφο κύριο Χίγκινς για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, το πρόγραμμα της Στοκχόλμη ορίζει ένα πλαίσιο για συνεργασία αστυνομική ε, τελωνίων, αστικού δικαίου, ασύλου, ε, μετανάστευση και πολιτική θεωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρουμε, το σχέδιο δράσης της Κομισιόν αναφέρεται στο πρόγραμμα στη Στοκχόλμη, το οποίο ε, εξετάζει σε έκθεσή τη η Επιτροπή Τζούρι. Υπάρχουν κάποιοι τομεί του σχεδίου δράση και του προγράμματο τη Στοκχόλμη που ε, άπτονται ε, τομέων ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Για παράδειγμα, τα πλαστά φάρμακα, τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, τα διανοητικά δικαιώματα και άλλα. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω Πιστεύω ότι η εναρμόνιση στην Ευρώπη θα είναι προ όφελο των ε, πολιτών και των εργαζομένων, αρκεί να γίνει με τρόπο δημογραφικό, δημοκρατικό και με τη μέθοδο των διαβουλεύσεων. Υπάρχουν πολλέ πτυχέ του προγράμματο τη Στοχόλμη που ανησυχούν ιδιαίτερα κάποιε οργανώσει ε, ε, πολιτικών δικαιωμάτων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δεν ε, πίπτουν στην ε, αρμοδιότητα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ε, να πω ότι κάποια πράγματα, με κάποια πράγματα δεν συμφωνώ. Το, να έχουμε ένα οχυρό Ευρώπη και άλλα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε μια συντονισμένη εκστρατεία κατά των ε, πλαστών προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών για να ε, διασφαλίσουμε την ε, προστασία των καταναλωτών και του ε, περιβάλλοντος. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι υπερβολικά τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε. Επίσης, όσον αφορά τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, καθότι απειλεί την υγεία των ανθρώπων. Ωστόσο πιστεύω ότι η εναρμόνιση των κανόνων ε, τελωνίου δεν θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να ε, απειλούνται τα γενώσιμα φάρμακα. Αυτή είναι μια ανησυχία που πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεσης βρίσκεται στους φακέλους σας. Ε, υπάρχουν παρατηρήσεις από άλλα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Γιακολίνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος σε αυτήν εδώ την πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων. Ε, άκουσα τον κύριο Higgins, ε, άκουσα την παρουσίαση όπως έγινε και θα ήθελα να πω όσον αφορά αυτή την ε, πρωτοβουλία θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ με το προλαλήσαντα συνάδελφο με απλώς κάποιες μικροδιορθώσεις θα έλεγα, μικρές αλλαγέ, ας πούμε. Εναρμόνιση. Εναρμόνιση είναι κάτι πολύ σημαντικό και γι' αυτό θεωρώ θα πρέπει εμείς να εκφραστούμε θετικά σε, αυτή την, σε αυτό το θέμα. Ακόμα και όταν έχουμε να, κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε θέματα που αφορούν και τα φάρμακα. Επίσης θα πρέπει κανείς να έχει σαφείς ορισμούς ξεκάθαρους και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να έχουμε έναν έλεγχο, ένα έλεγχο που λειτουργεί. Πολλές χώρες μέλη έχουν συζητήσει πάνω σε αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις δικές μας σχέσεις με τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα της Στοχόλμας ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φιλικό προς τον πολίτη. Μιλάει κανείς ε, για τα, τα δικαιώματα του πολίτη για να τέτοιο, μια τέτοια προσέγγιση και εμείς θέλουμε πραγματικά να έχουμε σαφέστατα ποια είναι τα όρια που υπάρχουν, ξεκάθαρες γραμμές. Για όσον αφορά δηλαδή το δικαίωμα ενός ατόμου και εγώ προσωπικά θα ήθελα να προτείνω κάποιες μικρές αλλαγές, αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, στην πρόταση. Με ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γιακολίνο από το ΕΛΚ. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος το λόγο, οπότε στρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος ή κυρία Σταμόιλεν, κάπως έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, καθορίζει το πλαίσιο για την προσεχή πενταετία στον τομέα της ε, δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Σημειώνουμε τις ανησυχίες και τα σημεία τα οποία ανέφερε ο εισηγητής για παράδειγμα σε σχέση με την παραποίηση καθώς και την ανάγκη να ε, παραμείνει η διάσταση του αστικού δικαίου κατά την εξέταση των σχετικών ζητημάτων. Σημειώνουμε επίσης την αναφορά στα δικαιώματα ε, των πολιτών, την ηθαγένεια που ενισχύεται η πτυχή αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει το σχέδιο δράσης το οποίο καλύπτει τα περισσότερα από τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν τα επόμενα πέντε χρόνια με στόχο την πρόθεση των στόχων ε, του προγράμματος της Στοκχόλμης. Επίσης θα υπάρξουν και άλλα μέτρα Δηλαδή θέλουμε να επικεντρωθεί το πρόγραμμα της Στοκόλμης στα μέτρα τα οποία θα ξεκινήσουν οι Γενικές Διευθύνσεις Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Δηλαδή δεν αποκλείουμε ορισμένα ζητήματα τα οποία έχετε θέσει να εμπίπτουν στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βέβαια θα αναφέρουμε τα σχετικά θέματα στους αρμόδιους υπαλλήλους των Γενικών Αυτών Διευθύνσεων που ασχολούνται με τα θέματα παραποίησης. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι η κατάθεση ε, τροπολογιών λίγη 28 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Α, ο κύριος... Ε, συγγνώμη. Ε, ναι, έχετε το λόγο. Δεν θέλω να καθυστερήσω, για ο κύριο Χίγκιν. Απλά θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τη γραμματεία τη Επιτροπής μα για τη βοήθεια που μου παρέσχει και για τον ε, συνήθω επαγγελματισμό που τη διακρίνει. Βέβαια, όπως είπατε, θα έχουμε τις τροπολογίες και θα τις μελετήσουμε. Thank you. Point four. Ευχαριστώ. Σημείο 4. Εμπορικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λατινική Αμερική. Συζητούμε το σχέδιο έκταση του Χέλμουτ Σόλτ από την ΚΟΕ. Νομίζω ότι έχουμε συζητήσει ήδη μία ή δύο φορές τουλάχιστον. Όπως ξέρετε, Κολομβία και Περού συνήψαν ε, στις αρχές του χρόνου ε, μάλλον ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις ε, και μετά και το Μάιο με την Κεντρική Αμερική και ολοκληρώθηκα συγκεκριμένα με την Κεντρική Αμερική. Επίση έχουμε με τον Μερκοσούρ συζητήσει ε, για τη σχέση σύνδεσης. Η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου φυσικά και θα παρακολουθεί του σύνεγγυ στις διαπραγματεύσει αυτέ. Εκτό από τι διαπραγματεύσει των εμπορικών συμφωνιών θα εξετάσουμε και το μελλοντικό πλαίσιο των εμπορικών μα σχέσεων με τη Λατινική Αμερική εν ώψη των δημόσιων διαβουλεύσεων που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελλοντική κατεύθυνση τη εμπορική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε και σχετική ανακοίνωση τον Οκτώβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον συνάδελφό μας Χέλμου Τσόλτση Σιγητή που θα μα ε, κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση. Uh, Έχετε νομίζω και στους φακέλους σας το σχέδιο έκθεσης. Χέλμουτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι πρώτη φορά που ασχολούμαστε τους τελευταίους μήνες με το θέμα αυτό. Θα ήθελα καταρχήν να ε, σας ευχαριστήσω ήδη για όσες ε, παρατηρήσεις ε, και προτάσεις ακούσαμε ε, κατά τη διάρκεια και της πρώτης παρουσίασης του εγγράφου και της πρώτης συζήτησης στην Επιτροπή μας. Στην έκθεση αυτή προσπάθησα να αναφέρω τα κύρια χαρακτηριστικά που διέπουν ε, το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με μια μεγάλη ήπειρο και να περιγράψω και τι μορφή θα μπορούσε να έχει το εμπόριο. Εξετάζουμε λοιπόν τις εμπορικές ε, σχέσεις ε, της ε, με την Λατινική Αμερική υπό το φως της γενικής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θέλω να το τονίσω ευθύς εξ αρχής. Πιστεύουμε ότι η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο του γενικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και κινούμαστε περισσότερο ε, προς την κατεύθυνση εταιρικών σχέσεων με τους ε, με τις ε, άλλες χώρες. Δηλαδή θέλουμε να συμπεριλάβουμε και πτυχές ε, οικονομικές, ε, απασχολησιακής πολιτικής, ε, περιβάλλοντος, οικονομικές, κοινωνικές κλπ. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία σύγχρονη στρατηγική εμπορική, εμπορική πολιτική Ε, που να υπαγορεύει τις κατευθύνσεις ε, για τους ε, αναγνωρισμένους εταίρους μας. Έτσι λοιπόν, ε, θέλουμε με αυτό να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων της ε, χιλιετίας του ΟΗΕ και θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ε, οικολογική βιωσιμότητα, την οικονομική ανάπτυξη. Είχαμε μία κρόαση για το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα για τις νέες προσπάθειες που γίνονται στην περιφέρεια αυτή για την διατήρηση της βιοπικιλότητας. Η βιωσιμότητα λοιπόν, η αηφορία αποτελεί σημαντική πτυχή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις εμπορικές σχέσεις. Τώρα που εκπονείται η μελλοντική εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε ως ε, ε, ευρωβουλευτές να συμβάλλουμε και εμείς. Πιστεύω ότι η χρονική στιγμή επόνησης αυτής της έκθεσης είναι πολύ καλή διότι εξετάζουμε τι ε, έχουμε καταφέρει με τις διαπραγματεύσεις, τι περιμένουμε στο μέλλον και πώς μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ε, συμφωνίες εμπορίου που έχουμε με την Λατινική Αμερική. εξετάζουμε και τις διαπραγματεύσεις Μερκοσούρ, βλέπουμε πώ όλες οι επιτυχίες αυτές ενσωματώνται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Αυτό έχω προσπαθήσει να δείξω στην έκθεσή μου αυτή. Τρίτον, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για το μέλλον της Λατινικής Αμερικής. Και να συμμετάσχουμε έτσι στην διαμόρφωση των εμπορικών μας σχέσεων. Προσπάθησα στην έκθεση να αναφέρω τις, τους ακρογωνιαίους λήθους μιας εμπορικής πολιτικής για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες μεγάλες περιφέρειες, με άλλες υπήρους. Προσπάθησα να μην χωρίσω την έκθεση στις επιμέρους εμπορικές συμφωνίες που υπάρχουν, αλλά να ακολουθήσω μια γενική κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύπλοκα τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το διπεριφερειακό εμπόριο. Εξετάζουμε λοιπόν το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Λατινική Αμερική γνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν με τη Συμφωνία Εμπορική Ένωσης Μεξικού, Ευρωπαϊκή ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κλπ. Γνωρίζουμε, έχουμε συζητήσει την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Κολομβία. Έχουμε λοιπόν εξετάσει τα επιμέρους θέματα. Πιστεύω όμως ότι σαν Επιτροπή έχουμε κοινή κατανόηση σχετικά με το τι μορφή θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει μια συμφωνία εμπορίου. Έχουμε συζητήσει για το πρόβλημα της μπανάνας. στα πλαίσια του ΠΟΕ και υπό το φως των νέων συμφωνιών με το ε, Περού και την Κολομβία. Όταν μιλάμε για τη μελλοντική εμπορική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Λατινικής Αμερικής, θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι η ε, ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών της Λατινικής Αμερικής ε, είναι σημαντική για την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εμπορικό εταίρο. Χώρες όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Κολομβία, το Περού ε, θα πρέπει να εξεταστούν. Επίσης, θα πρέπει τα πολύπλοκα ζητήματα που ανέφερα να δούμε πώς μπορούμε να τα λύσουμε στα πλαίσια των εταιρικών μας σχέσεων με τις χώρες αυτές, των μεγάλων και των μικρών χωρών. η απασχόληση στη Λατινική Αμερική, η θέση απασχόληση στη Λατινική Αμερική, η ανάπτυξη των οικονομιών ε, αποτελούν ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα είναι προς αμοιβαίο συμφέρον. Κατά την αιτιολόγηση της νομοδότησής μου προσπάθησα να απαριθμίσω τα θέματα αυτά. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Κλείνοντας ε, θα ήθελα να πω ότι φυσικά ως εισηγητή πρέπει να προσέξω η έκθεσή μου ε, να, μην είναι, να μην περιέχει παραπάνω από 12.000 ε, χαρακτήρες. Γι' αυτό αναγκαστικά περιορίστηκα. Προσπαθώ όμως ε, να έχω στο, σε όλη μου την έκθεση αυτό το συνδετικό νήμα. Βλέπω στην ανταλλαγή απόψεων, στη συζήτηση της έκθεσής μου, διότι έτσι μπορεί να έχω την ευκαιρία να ξανασκεφτώ ενδεχομένως κάποιες πτυχές, ε, να υποβάλω τροπολογίες. Η προθεσμία έχει τεθεί στο τέλος του Ιουλίου. Λίγες μέρες ε, δηλαδή πριν φύγουμε όλοι για διακοπές ε, θα έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα στο τέλος του καλοκαιριού, αρχή του φθινοπόρου, να συναντηθούμε σε ομάδα εργασίας, να εξετάσουμε τις τροπολογίες, ώστε το αποτέλεσμα να είναι μία έκθεση με στόχο την διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τη Λατινική Αμερική για τα επόμενα δέκα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χέλμουτ Σόλτς. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. ο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλτ για την έκθεσή του που θεωρώ ότι είναι μια έκθεση που πηγαίνει προ σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ και εγώ ότι η Λατινική Αμερική είναι ένας από τους βασικούς μας εταίρους και σε αυτές τις ε, στιγμές κρίσης νομίζω ότι θα πρέπει να συμπήξουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την περιοχή αυτή γιατί αυτό θα βοηθήσει γενικότερα ένθερκα κύθνο του Ατλαντικού. Θεωρώ επίσης ότι είναι και μια ευκαιρία για να εξαγάγουμε και τις ευρωπαϊκές αξίες ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινωνικές πτυχές αλλά και άλλες πτυχές όπως ε, οι σχετικές με το περιβάλλον. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλά μπορεί, αλλά και οφείλει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στη Λατινοαμερικανική Ήπειρο. Θα ήθελα παρόλα αυτά να επισημάνω κάποιες μικρές διαφορές, αν θέλετε αποκλήσεις ε, προσωπικές σε σχέση με τα όσα λέει ο ηγετής. Παραδείγματος χάρη. Ο κίνδυνος ε, συμφωνιών ε, σε διαφορετικές ταχύτητες, στην σκέψη H, λατινικό. Σε ό,τι αφορά την Κεντρική Αμερική, ξέρουμε ότι η σχετική συμφωνία είχε ω επίκεντρο τη συμφωνία περιοχή προ περιοχή. Ενώ στην, στην περίπτωση Κολομβία-Περού πρόκειται για επέκταση ε, τη συμφωνία σύνθεση με όλη την κοινότητα των Άνδεων. Εμείς πιστεύω ότι δεν ε, υπάρχει οποιαδήποτε αποσύνθεση ή αποδιάρθρωση, αλλά αντίθετα σύνδεση, μεγαλύτερη σύνδεση ε, των χωρών αυτών που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παράγραφο 18 γίνονται κάποια αναφορές. Ε, ε, στόχος... Ε, νομίζω ότι θα, θα πρέπει η ομάδα μας να μην δημιουργήσει καμία τροχοπέδη σε καμία χώρα η οποία θα θέλει να προχωρήσει. Στις 4 Ιουνίου επίσης η κυβέρνηση της Βολιβίας δήλωσε ότι προτίθεται να αποσύρει το αίτημα το οποίο είχε υποβάλει στο δικαστήριο και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την οικονομία των λατινοαμερικανικών χωρών, ότι βασίζεται σε τομεί μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Εμεί θεωρούμε ότι η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων θα βοηθήσει στη μείωση των ανισορροπιών που ενδεχομένω υπάρχουν και θα προσελκύσει επενδύσει σε πιο παραγωγικού τομεί στην περιοχή αυτή. Θέλουμε επίση να τονίσουμε τη σημασία του ότι οι χώρε της Λατινικής θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξουν και εσωτερικέ διαρθρωτικέ κοινωνικέ φορολογικέ μεταρρυθμίσει που θα συνοδεύουν αυτέ τι συμφωνίε ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία. Ο εισηγητή επίση στην παράγραφο 25 μιλά και για το νέο μηχανισμό επενδύσεων και τη σημασία του στη Λατινική Αμερική. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τη σημασία που έχει ο μηχανισμό αυτό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που είναι και αυτές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Θέλω να ευχαριστήσω κατά κλείδι τον κύριο Σόλτ για την προσπάθειά του να του πω ότι θα καταθέσουμε τροπολογίε ε, για να ληφθεί υπόψη ε, ε, η διαφοροποίησή μα σε αυτά τα σημεία τα οποία ανέφερα πριν και βέβαια να του δηλώσω ότι θα είμαστε στη διάθεσή του για οποιαδήποτε συνεργασία. Ευχαριστώ. Εμίλιο Μενέντεθ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, προσπάθεια που εφιέρωσε ο συνάδελφος Σόλτς νομίζω ότι παίρνει σάρκα και οστά στην έκθεση αυτή και πρέπει να τον συγχαρούμε για την έκθεση. Είδαμε ποια είναι η βασική ιδέα που διατρέχει την έκθεσή του Μπορεί να διαφωνούμε ενδεχομένω με κάποια σημεία, αλλά νομίζω ότι η έκθεσή του παρόλα αυτά είναι συνεπής και συνεκτική. όπως και ο προλαλής σας, και εγώ θεωρώ ότι στόχος μας είναι να εξαγάγουμε τις αξίες μας στη Λατινική Αμερική και υπάρχει, ε, όχι ψύχο, τέλο πάντων, μια σημασία, αν θέλετε, που δίνει ε, σε αυτήν την ομάδα εργασία ο κύριο Σόλτ. Εντάξει, συμφωνούμε όλοι, αλλά θα πρέπει να είναι συμβατή και με τι αξίε μα αφενός και με τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφετέρου. Δηλαδή, να γίνουν κατανοητές οι αξίες και τα συμφέροντα βέβαια θα υπόκεινται και στον δέοντα έλεγχο και δεν θα πρέπει να υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ αυτών. Φυσικά ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στη Λατινική Αμερική όσο και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη είναι επίση προτεραιότητα που με βρίσκει σύμφωνο. Τούτων λεχθέντων, δεν θέλω βέβαια να μακρηγορήσω γιατί και εγώ θα καταθέσω τροπολογίε, θέλω πάντως να κάνω κάποιε σύντομε παρατηρήσει. Στην παράγραφο ε, ο συνάδελφος ε, Σόλτ, λέει ότι το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής είναι ασυμμετρικό. Εγώ πρέπει να πω ότι θα έπρεπε να λέμε με ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όχι με όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, γιατί αυτό αφήνει να ιονιθεί η διατύπωση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Στην παράγραφο 6, ο εισηγητής λέει ότι χαιρετίζει τις εξελίξεις στην Βραζιλία, τον Ισημερινό και τη Βολιβία. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερο γιατί μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για τις χώρες αυτές για να καταλάβουμε την κατάσταση στη Λατινική Αμερική, να βάλουμε από τη μία τη Βραζιλία και από την άλλη τον Ισημερινό και τη Βολιβία. Εγώ θα έλεγα όμω ότι την ανάπτυξη νέων εμπορικών πολιτικών και πολιτικών στον τομέα των πόρων έχουν οδηγήσει στην, στον περιορισμό τη φτώχεια και των ανισοτήτων και να μην κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση και να μην μιλήσουμε για Βραζιλία, Ισημερινό και Βολιβία. Η παράγραφος 15 τώρα με κάθε σεβασμό προς τον εισηγητή είναι λίγο πατερναλιστική ως προς τη διατύπωσή της. Εγώ δεν νομίζω ότι η Κομισιόν ή η Ευρώπη μπορεί να θεσπίσει αποτελεσματικό μηχανισμό καταγγελιών για τη Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι η ίδια η Λατινική Αμερική είναι αυτή που θα πρέπει να θεσπίσει το σχετικό μηχανισμό. Το λέω με κάθε σεβασμό βέβαια. Ε, είναι παράλογο να ζητούμε εμείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θεσπίσει στη Λατινική Αμερική ένα μηχανισμό είναι ένας ε, έτσι ήπιος τρόπος ε, να τους δώσουμε κατευθύνσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά του δασμού ε, για την μπανάνα, στο σημείο 16 δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχουν τόσε πια διαφορέ, νομίζω ότι έχουν επιληθεί. Εν γέννη, έτσι, εν γέννη. Παράγραφο 17. Έχουμε ένα πρόβλημα ερμηνεία. Στα αγγλικά και στα ισπανικά, στο 17 οι δύο γλωσσικές εκδοχές διαφέρουν, όχι δραματικά, αλλά διαφέρουν. Δεν ξέρω τι λένε τα γερμανικά, αλλά στα αγγλικά, στο σημείο 17, λέει stresses that parliaments still have to ratify the agreement. Στα ισπανικά λέει ορισμένα κοινοβούλια πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία. Δηλαδή, στα αγγλικά λέει τα κοινοβούλια, τονίζω ότι τα κοινοβούλια δεν έχουν ακόμα επικυρώσει, ενώ στα ισπανικά λέει ορισμένα κοινοβούλια δεν έχουν επικυρώσει. Νομίζω ότι πρέπει να τροποποιηθεί η φράση αυτή. Είναι προφανέ ότι πρέπει να επικυρώσουν τη συμφωνία τα κοινοβούλια. Ε, είναι σαν να λέμε ότι η Κομισιόν έχει νομοθετική πρωτοβουλία. Ε, δηλαδή λέμε κάτι αυτονόητο. Φυσικά και πρέπει τα κοινοβούλια να επικυρώσουν. Και ολοκληρώνω ότι θα αποσύρει ε, αυτό το, το αίτημα ε, στο δικαστήριο, στο Διεθνές Δικαστήριο. Το έχω ξαναπεί, νομίζω και εγώ ότι πρέπει να διαγραφεί αυτό το σημείο. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης τη διαπραγματευτικής εντολής κτλ. κτλ. Εγώ νομίζω, και η ομάδα μου το ίδιο πιστεύει, ότι ο Επίτροπος ε, Ντεχούχτ τα έχει πει και αυτός. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ε, πούμε με τα λόγια αυτά. Άλλο να πούμε ότι πρέπει να τονίσουν περιοδικές μελέτες ε, εξολόγησης επιπτώσεων. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Να το πούμε έτσι. Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει την Σουρ και εμείς να την επενέσουμε, αλλά και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί λέει ο ότι τονίζει το ρόλο τη Ουνασούρ, τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει στο μέλλον. Όχι, ήδη διαδραματίζει ο UNASUR ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα θυμάστε ότι με πρωτοβουλία της Βραζιλίας, πριν κάποιο καιρό, η UNASUR, η Ένωση δηλαδή των Εθνών της Νοτιού Αμερικής, απέτρεψε μια εμπόλεμη σύραξη. Παραλαμβάνω πρωτοβουλία της Βραζιλία. Να βάζουμε λοιπόν θα μπορούσε να διαδραματίσει ήδη, να το βάλουμε στον ενεστώτα, ήδη διαδραματίζει. Ο συνάδελφος Στάλβα και όλοι οι άλλοι βέβαια συνάδελφοι ως ε, αλληλέγγυοι Ευρωπαίοι πολίτες νομίζω θα στηρίξετε την αναφορά στις επιτυχίε τη Ισπανική Προεδρία όπως θέλουμε στο διατυπώσουμε, αλλά νομίζω ότι η διάσκεψη κορυφής της Μαδρίτης έδωσε μια όθηση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Στέβη, αντιπρόεδρός μας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σόλς, θα είναι δύσκολη η μάχη. Αναφέρατε και θα ήθελα να σχολιάσετε ένα σημείο εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημείο 19 στη σελίδα 8 λέει ο μιλητής. Αναφέρεται στην ε, Λέει ότι τονίζει ότι πρέπει να συμμετάσχει από κοντά σε όλα τα βήματα των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ. Ερώτηση. Έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με την Μερκοσούρ από τότε που ε, συζητούσαμε το DDA. Και δεύτερον, εσεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να απαντήσετε ε, τι ερωτήσει σχετικά με την Αργεντινή και το μπλοκάρισμα των μεταποιημένων επεξεργασμένων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασμένων προϊόντων που προέρχονται από τη Βραζιλία. Η Mercosur πρόκειται να διευρυνθεί, φαίνεται όμως να υπάρχει αρκετή ανησυχία εντός της ομάδας Mercosur. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή προς τον κύριο Σόλς. Ο, ο κύριος Πάρτμοθ. Εκτός μικροφώνου δεν ακούμε. Ζητώ συγγνώμη. Τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω πολύ σύντομα. Πρώτον, είναι εξαιρετική η έκθεση αυτή. σύμφωνα και με τα πολύ απαιτητικά κριτήρια του, της Ευρωπαϊκής και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και τους αδέρφους του που εκπώνησε μια τόσο ε, εύληπτη έκθεση. Ε, δεν θα σας εκπλήξει το ότι δεν συμφωνώ με όλα αυτά όμως και ιδιαίτερα με απασχολεί η παράγραφος 1 που λέει ότι επισημαίνει ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα ορίζει την εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω αναπόσπαστο τμήμα τη συνολική εξωτερική δράση τη Ένωση. Θα ήθελα εκ μέρου ε, του κόμματό μου και τη πολιτική μου ομάδα να πω ότι πιστεύουμε ότι το εμπόριο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο, δεν θα πρέπει να ε, αποτελεί αντικείμενο πολιτικών ε, προγραμμάτων. Θα δυσκολευτούμε λοιπόν πολύ να συμφωνήσουμε με την παράγραφο 1. Ε, κατά τα άλλα προσλέπω στην εμβάθυνση στο θέμα αυτό, στις άλλες ευκαιρίες συζήτησης που θα έχουμε. Απλά ήθελα να κλείσω όπως ξεκίνησα συγχαίροντας τον εισηγητή για μια εξαιρετικά καλογραμμένη έκθεση που θα αποτελέσει εξαιρετική βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ. Σημειώνουμε τον έπαινό σας. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ματίας Γιώργενσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, ε, θα κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Θα επαναλάβω κάποιες γενικές παρατηρήσεις που έκανα την προηγούμενη φορά. Δεν θα επαναλάβω μάλλον τις παρατηρήσεις που έκανα την προηγούμενη φορά, απλά να πω ότι συμφωνούμε απόλυτα ότι θα πρέπει να έχουμε μία συνεπή θέση ως προς το εμπόριο μας με την ε, Λατινική Αμερική, το οποίο να επιδιώκει και τους γενικότερους στόχους της κοινωνικής συνοχής και της ε, περιφερειακής ε, ολοκλήρωσης. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Λατινική Αμερική επιδιώκει όχι να έχει μία μακροπρόθεσμη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, αλλά να έχει κάποιες πιο βραχυπρόθεσμες συμφωνίες, οι οποίες όμως να ενσωματώνουν και τον πολιτικό διάλογο, ε, άλλε δραστηριότητες και την ε, χρήση επιδοτήσεων. Σε σχέση με αυτά που κάνουμε με τη Λατινική Αμερική για τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ή συμφωνίες, συμφωνίες σύνδεσης, Όλα αυτά είναι απόλυτα ε, ε, συνεπή με αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΠΟΕ. Γενικά, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, ε, παρακολουθούμε την δουλειά που συνεχίζει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα αυτών και περιμένουμε με ανυπομονησία την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Για τον σημαντικό αυτό τομέα στις στη δουλειά μας για την εξωτερική πολιτική και την εμπορική πολιτική. Όπως είδατε με τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει πρόσφατα, κάποιες από τις προσπάθειές μας ε, φέρουν καρπούς. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα να απαντήσω και στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Όσον αφορά τα προβλήματα των εισαγωγών ε, ευρωπαϊκών τροφίμων στην Αργεντινή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε πάρει πολύ στα σοβαρά. Έχουμε συζητήσει το θέμα μέσω διπλωματικών καναλιών εδώ στις Βρυξέλλες. Έχουμε κάνει επίσημα διαβήματα στην Αργεντινή. Σε ε, επίσημο επίπεδο έχουμε ε, θίξει το θέμα απέναντι στις, ε, ε, στις αρχές της Αργεντινής σε εκδήλωση που έγινε πριν δύο εβδομάδες στο Buenos Aires και το αναφέραμε αυτό και στην επίσημη συνάντηση όπου είχαν προσληθεί όλοι οι εταίροι Μερκοσούρ της Αργεντινής για να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις της αντιπροσωπείας μας δείχνουν ότι έχουν κάποιο αποτέλεσμα οι προσπάθειες και ότι τα κοντέινερ ευρωπαϊκής προέλευσης που είχαν μπλοκαριστεί φαίνεται να ξεμπλοκάρονται τώρα. Δεν έχουμε ακούσει νέες περιπτώσεις που να έχουν οδηγήσει σε προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να πούμε ότι οι ενέργειές μας είχαν αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε όμως να εξετάζουμε σοβαρά το θέμα και θα συνεχίσουμε να το επισημαίνουμε απέναντι στην Αργεντινή και τους εταίρους μας στην Mercosur. Ναι, η Μερκοσούρ διευρύνεται. Πρόκειται για την ελευθερία των μηχανισμών ε, περιφερειακή ολοκλήρωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε διευρύνεται. Όταν λαμβάνουμε σχετικέ αποφάσει, δεν επιτρέπουμε σε άλλου εταίρους να ε, επηρεάσουν τι αποφάσει μα. Είναι λοιπόν δικαίωμα της Μερκοσούρ να διευρυνθεί όσο θέλει. Η διεύρυνση με τη Βενεζουέλα προχωράει πολύ αργά, περιμένει ακόμα επικύρωση στο Κοινοβούλιο της Παραγουάης και κατόπιν θα ακολουθήσει μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία ε, κατά την οποία θα πρέπει η Βενεζουέλα να υιοθετήσει το κεκτημένο της Μερκοσούρ. Τώρα το πότε λοιπόν πώς, ε, και πώς η Βενεζουέλα θα καθίσει στο τραπέζι σαν ε, ισότιμος εταίρος, ως ισότιμος εταίρος, αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν, συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ο κύριος Σούλς, ε, Σόλς να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσο γίνεται πιο σύντομα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και για την εκτίμησή τους για τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα πάνω στην έκθεση αυτή. μία παρατήρηση. Άκουσα και την νέα. Ε, μία απάντηση προς τον συνάδελφο. Εμπόριο και ε, εξωτερική πολιτική. Ε, το εμπόριο, η, εξωτερική, η εμπορική πολιτική είναι μία πτυχή των εξωτερικών μας δράσεων και εκτιμάται ως τέτοια, κρίνεται ως τέτοια, καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, να ενεργεί ως φορέας ε, στις εξωτερικές αυτές δράσεις. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ο εξωτερικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν φαίνεται εδώ και ε, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των διαφόρων τομέων. Αυτό είναι μια σκέψη ε, που θα, πρέπει να έχουμε κατά νου κατά την διαμόρφωση του εξωτερικού εμπορίου στο μέλλον και ε, απέναντι στη Λατινική Αμερική. Όσον αφορά την Μερκοσούρ, θα ε, μπορούσα μόνο να συμφωνήσω με την Κομισιόν. Το πώς αναπτύσσεται η Μερκοσούρ είναι θέμα των χωρών αυτών. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εκεί που θα επηρεάσει τις μελλοντικέ σχέσεις ε, χωρών Μερκοσούρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας κατά, το, ε, ε κατά τις εμπορικές μας σχέσεις με την περιφέρεια αυτή. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα μελλοντικά μας βήματα μπορεί να τα διατυπώσει κανείς αυτά με ε, διάφορους τρόπους. Πολλά από αυτά τα πράγματα ισχύουν όχι μόνο για μία χώρα, αλλά επηρεάζουν το χαρακτήρα των μελλοντικών σχέσεων εμπορικής, ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής γενικά. Όσον αφορά το σημείο 17, νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα σε το αγγλικό κείμενο είναι όμοιο με το γερμανικό. Θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συνεργάς την ε, κυρία Πρίπας και για την πολύ αντικειμενική ε, συνεργασία της στην έκθεση αυτή. ως εισηγητής μπόρεσα να συμμετάσχω σε διάφορες αντιπροσωπείες ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα αυτή. Ευχαριστώ να επενθυμίσω για να κλείσουμε το θέμα αυτό ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 28 Ιουλίου το μεσημέρι και Πριν προχωρήσω στο σημείο 5. Α, για την ώρα. 6 με διορθώνουν. 6 ώρα είναι η λήξη προθεσμίας. 28 Ιουλίου. Το απόγευμα φυσικά. Έχει διανεμηθεί το δελτίο μου στο Περθμόν 4 και θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία που προετοίμασαν όλες αυτές τις ε, πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, Βλέπω ότι αφήχθη ήδη ο προσκεκλημένο μας. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 6 της ημερησιάς διάταξης. Να καλωσορίσω τον κύριο Στίβεν Βανάκερε, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Υπουργό Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου στην βελική κυβέρνηση. Ο κύριος Βανέκερε εκπροσωπεί την Προεδρία του Συμβουλίου για το τρέχον εξάμεινο. Βρίσκεται εδώ για να μας αναφέρει τις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. μετά από την επιτυχή Ισπανική Προεδρία. Τώρα λοιπόν να τη σκητάλη παίρνει το Βέλγιο για την εκπεριτροπής Προεδρία και προσβλέπουμε σε μια εξίσου επιτυχημένη Προεδρία με τις προηγούμενες. Σας εύχομαι καλή τύχη λοιπόν κύριε Βανάκερε και σε εσά προσωπικά και στην κυβέρνησή σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλώς ορίσατε για μια ακόμη φορά και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω για τα γενικά σας λόγια, ε, για το καλωσόρισμα. Τα λόγια σας μου δίνουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να, να υπογραμμίσω κάτι που πάντοτε ε, λέγαμε και τονίσαμε και παρουσιάζοντα τι προτεραιότητέ μα στο Στρασβούργο. Δηλαδή ότι θέλουμε να έχουμε καλή σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιλαμβανόμαστε πλήρω τον όλο και αυξανόμενο και σημαντικότερο ρόλο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη θέση και τη συνθήκη τη Λισαβόνα και θα το λάβουμε αυτό υπόψη μα. Και είναι σαφέ ότι και αν δει κανεί ε, τη διάταξη του Συμβουλίου, το σχηματισμό δηλαδή του Διεθνούς Εμπορίου, λαμβάνουμε υπόψη μας ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι προτεραιότητες που θα σας παρουσιάσω θα πρέπει βέβαια να εδωθούν, ε, ως, να εννοηθούν μάλλον ως τμήμα της πρότασης της Τρόικας Ισπανίας, Βελγίου, Ουγγαρίας όπως ε, ο Ισπανός συνάδελφος στις 23 Ιουνίου σας παρέ, παρουσίασε την πρόοδο του έργου του Συμβουλίου για το πρώτο εξάμεινο, εγώ ελπίζω με την πλευρά, από την πλευρά μου ότι θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο για την εκπλήρωση των στόχων που έχουμε αναλάβει λαμβάνοντα βέβαια υπόψη το πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν, τι διαπραγματεύσει που είναι σε εξέλιξη αλλά και τι αλλαγέ που έχει επιφέρει η συνθήκη τη Λισαβόνα και επί τη ουσία και σε ό,τι αφορά τι νέε αρμοδιότητε των, θεσμικών οργάνων. Ω γενική παρατήρηση νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να σα υπενθυμίσω το μέγεθο τη κρίση που βιώσαμε και εξακολουθούμε να βιώνουμε στην Ευρώπη και ότι θα πρέπει βέβαια να εξεύρουμε βιώσιμε λύσει βασισμένε στην ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κοινή εμπορική πολιτική σίγουρα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα τη οικονομική μεγέθυνση και τη απασχόληση. Δεν είναι βέβαια πανάκια, σίγουρα όμω θεωρούμε ότι είναι ένα τμήμα της λύσης. Εάν μαζί με όλα τα κράτη-μέλη και τα 27 καταφέρουμε να δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να επιβεβαιώσουμε και να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας ε, προς όφελος των πολιτών μας και να υποστηρίξουμε όμως ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη και των φτωχότερων χωρών. Σε ό,τι αφορά τους στόχους μας, σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου, είμαστε υπέρ ε, της πολυμερούς προσέγγιση Θα σας μιλήσω για τη νέα διαδικασία της Συνθήκης τη Λισαβόνας και τι επιπτώσεις έχει αυτή για την εξισορρόπηση μεταξύ, την ισορροπία μάλλον μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Θα σας μιλήσω επίσης ε, για τις εμπορικές μας σχέσεις με τους κύριους ε, εταίρους. Θα σας μιλήσω για την αναπτυξιακή διάσταση του εμπορίου και εν τέλει θα σας μιλήσω για, την, ε, το θεματολόγιο της Ελληνικής Προεδρίας και την ΑΚΤΑ. Έτσι λίγο πολύ να σας δώσω το σκελετό της παρουσίασης μου. ό,τι αφορά την πολυμερή προσέγγιση λοιπόν για την απελευθέρωση του εμπόριου όπως σας είπα, είμαστε ως Βελική Προεδρία υπέρ αυτής της πολυμερούς ε, προσέγγισης και διαδικασίας. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν νομίζω ότι προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα παραμένει στο, ε, στο, στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Γνωρίζετε ποια είναι η ευρωπαϊκή θέση. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε κάποια ζητήματα αυτή την στιγμή με το χρονοδιάγραμμα, αλλά η συμφωνία νομίζω ότι θα δώσει μεγάλη όθηση στην παγκόσμια οικονομία, ιδίω για τι αναπτυσσόμενες χώρε και θα συμβάλλει στην πρόληψη κάποιων ε, τάσεων ε, προστατευτισμού. Ε, βέβαια δεν μπορεί μόνη της Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τη διαφορά. Τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής της ομάδας των 20 στο Τωρόντο στο τέλος του Ιουνίου νομίζω ότι μας συνιστούν να είμαστε ρεαλιστές ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και αν υπάρξουν νέε εξελίξεις σίγουρα η Προεδρία μαζί με την Επιτροπή θα ενημερώσουν το Κοινοβούλιο όπω συνέβη μέχρι τώρα και όπως άλλωστε επιτάσσει και η συνθήκη. Όταν τώρα μιλάμε για τη διαπραγμάτευση περιφερειακών και δημερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Θέλω να τονίσω ένα σημείο. Ποτέ στόχο μα δεν θα είναι να αντικατασταθεί το πρώτο κεφάλαιο, δηλαδή οι πολυμερεί συμφωνίε. Δεν είναι αυτό ο στόχο. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, πράγματι οι περιφερειακές και οι διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ολοκληρώνουν την επεωρική απελευθέρωση που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης των ΠΟΕ και βοηθούν ε, να γίνουν κάποιες διευθετήσεις για ζητήματα που δεν αποτελούν αντικείμενο των συζητήσεων του ΠΟΕ. Η Προεδρία μας λοιπόν θα εργαστεί για να επιτευχθεί η πρόοδος της ε, διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη σε περιφερειακό επίπεδο με τη Euromed, με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, με τη Mercosur, αλλά και σε διμερές επίπεδο με χώρες όπως Ινδία, Σιγκαπούρη, Καναδάς, Ουκρανία. Και όπου είναι δυνατόν ο στόχος μας θα είναι η ολοκλήρωση των συμφωνιών. Θα ήθελα να επικεντρωθώ καταρχά στι περιφερειακέ διαπραγματεύσει. Πρέπει να πω ότι γνωρίζω τις ιδιαίτερότητε ε, τη κάθε μια ξεχωριστά από τι περιφερειακέ διαπραγματεύσει. και το γεγονό επίση ότι πολλέ από αυτέ ή συνεχίζουν για χρόνια ή διεκόπησαν, ενεστάλησαν για κάποια χρόνια. Αυτά τα γνωρίζω. Όταν λοιπόν αξιολογούμε το δυναμικό ολοκλήρωση σύναυση των συμφωνιών αυτών θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα όλα τα στοιχεία όπω λαμβάνουμε βέβαια υπόψη μα και τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών. Θα παρακολουθούμε λοιπόν ως Συμβούλιο από κοντά τις εξελίξεις βάσει των εκθέσεων της Κομισιόν και έχοντας υπόψη μας ε, τους όρους και τις προϋποθέσεις ε, που ορίζονται από τις ε, οδηγίες μας για τις διαπραγματεύσεις. Για να είναι επιτυχημένη η συμφωνία με την Μερκοσού παραδείγματο χάρη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές Παραδείγματο χάρη, βιομηχανικά αγαθά, υπηρεσίε, γεωργία αλλά και προστασία δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία ε, και κυβερνητικέ δημόσιε συμβάσει. Σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει τη Euromed, γνωρίζετε ότι ο στόχο μα είναι ένα χώρο ελεύθερων συναλλαγών που θα προβλέπει την προοδευτική απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη τη περιοχή και θα συμπεριλαμβάνει νομικά δεσμευτικέ διατάξει στον τομέα του εμπορίου και τη οικονομική ρύθμιση. Θα ξέρετε επίση ότι στα τέλη του προηγούμενου έτου θεσπίσαμε και έναν οδικό χάρτη για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή πέραν του 2010. Και με την Επιτροπή και τους άλλους μας εταίρους θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης. Σε ό,τι αφορά την Κεντρική Αμερική, το Συμβούλιο δεν έχει την επίσημη πρόταση της Κομισιόν για υπογραφή της συμφωνίας που ολοκληρώθηκε το Μάιο. Θα υιοθετήσει λοιπόν το ε, Συμβούλιο την απόφαση σύναψης της συμφωνίας αφού θα έχει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 218 παράγραφος 6, σημείο α της συνθήκης. Και σε ό,τι αφορά τώρα τι διαπραγματεύσει ε, με το Συμβούλιο Συνεργασία του Κόλπ και παρά την πρόοδο που έχουμε σε διάφορα θέματα, παραμένουν ανεπίλητα κάποια ζητήματα όπω το εμπόριο. Και ένα κοινό ε, συμβούλιο που πρόσφατα συνήλθε για την 20η φορά συζήτησε τα ζητήματα των εξαγωγικών δασμών. Όλες τις θετικές εξελίξεις θα τις παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Έρχομαι τώρα στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Ε, δεν είναι ούτε αυτό απορίας άξιων. Ε, ολοκληρώνεται η συμφωνία μας με την Νότια Κορέα. Αυτή είναι, μάλλον η ολοκλήρωση της συμφωνίας μας είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή συζητούμε μαζί σας τη ρήτρα διασφάλισης. Η διαδικασία που οδήγησε στην απόφαση υπογραφής και προσωρινή εφαρμογή τη συμφωνία έχει ήδη ξεκινήσει αφού ε, αποφάνθηκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρόκειται για την πιο φιλόδοξη συμφωνία που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2006 η στρατηγική μας Global Europe το γνωρίζει το Συμβούλιο, γνωρίζει και την ανάγκη εξολόγηση τη συμφωνία και όλων των πολιτικών και οικονομικών διαστάσεων και πτυχών τη για να υπάρξει μια εξισορρόπηση μεταξύ των συμφερόντων μα αλλά και τη αποτελεσματικότητα τη ρήτρα διασφάλιση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να έχει το τελικό κείμενο τη συμφωνία στη διάθεσή του μετά το καλοκαίρι για να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Επίση, θα θυμάστε ότι η διαδικασία διαπραγμάτευση συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών ΑΣΕΑΝ αποδείχθηκε ιδιαίτερα βραδία και δύσκολη. Σταμάτησαν λοιπόν οι περιφερειακές συνομιλίες κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών για να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την διμερή διαδικασία με τις ενδιαφερόμενες χώρες, έχοντας όμως στο μυαλό μας για πιο μακροπρόθεσμα βέβαια και το ενδεχόμενο περιφερειακή συμφωνία. Αυτές λοιπόν οι συμφωνίες ε, οι διμερείς θα αποτελούν ε, ε, τα λιθαράκια τα οποία στη συνέχεια θα συγκροτήσουν με μια περιφερειακή συμφωνία. Με τη Σιγκαπούρη ήδη έχουν γίνει δύο γύροι διαπραγματεύσεων το 2010 και προβλέπεται ένας τρίτος για το Σεπτέμβριο διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδία ξεκίνησαν το 2007 και μέχρι στιγμής έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις που μας έδωσαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις προσδοκίες των πλευρών. Έχει υπάρξει πρόοδο, υπάρχουν όμω κάποιοι ακαθόδει τομεί όπω είναι οι δασμοί και τα ζητήματα των συμβάσεων, των προμηθειών. Ελπίζουμε να υπάρξει σημαντική πρόοδο στι διαπραγματεύσει ε, στη διάρκεια του παρόντο έτου, αλλά μάλλον δύσκολο είναι να προβλέψει κανεί ε, ε, την έκβαση για φέτος. Τώρα με τον Καναδά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαπραγματεύεται μια συνολική οικονομική εμπορική συμφωνία, ΣΥΤΑ, ΣΕΤΑ, δηλαδή μια ευρεία συμφωνία η οποία θα εμβαθύνει τις οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις. Πρόκειται για μια φιλόδοξη πρωτοβουλία, η οποία ε, απορρέει από μια κοινή διερευνητική άσκηση που θα καλύπτει τα ενδεχόμενα ωφέλη και για τις δύο πλευρές σε τομεί όπω είναι τα αγαθά, υπηρεσίε, οι δημόσιες συμβάσεις, προστασία, εφαρμογή των δικαιωμάτων ε, πνευματική ιδιοκτησία, δεσμεύσει για τι κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ πτυχέ, εμπορίου και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα πράγματα προ τη σωστή κατεύθυνση και να μπορέσουμε να κάνουμε μια απογραφή τη κατάσταση των το φθινόπωρο για να δούμε αν είμαστε στο ίδιο μήκος και αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η Ουκρανία τώρα είναι στην μέρη διάταξη από το 2008. Ένα γύρο διαπραγματεύσεων έχει ήδη λάβει χώρα. Η πρόοδο φαίνεται όμω εν γέννη δύσκολη στην παρούσα φάση, ιδίω ό,τι αφορά ζητήματα για την ρυθμιστική προσέγγιση και την πρόσβαση στην αγορά για ορισμένου τομεί. Η Ουκρανία πάντω είναι ένα σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο ελπίζει να προχωρήσουν στο επόμενο εξάμεινο και οι διαπραγματεύσει. Εν τέλει να αναφέρω τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με το Περού και την Κολομβία. Αφού η Κομισιόν ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την πολυμερή συμφωνία το Μάρτιο του 2010, Περιμένει τώρα τις επίσημες προτάσεις της Κομισιόν για να ξεκινήσει η διαδικασία υπογραφής και σύναψης της συμφωνίας. Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι ολοκληρώνω το τμήμα που αφορούσε τις διμερείς ε, διαδικασίες και διαπραγματεύσεις. Τώρα, σε ένα τρίτο κεφάλαιο θα ήθελα να επισέλθω σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, που όπως γνωρίζετε επέφερε μείζονε αλλαγές στην κοινή εμπορική πολιτική. Μια από αυτές, πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, αφορά τη μεγαλύτερη αρμοδιότητα, την αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση εσωτερικών μέτρων για την υλοποίηση της κοινή εμπορικής πολιτικής, καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Προβλέπει επίσης ε, η συνθήκη την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κοινοβούλιο. Εμείς ως Προεδρία χαιρετίζουμε τις σημαντικές αυτές αλλαγές και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ε, αναγνωρίζουμε και διαπιστώνουμε ότι ξεκίνησε ήδη αυτή η στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εμπορικά θέματα. Και εμεί θα φροντίσουμε να εφαρμοστούν πλήρω οι διαδικασίε τη συνθήκη τη Λισαβόνα σύμφωνα με του στόχου τη εμπορική πολιτική τη Ένωση. Μια μείζων αλλαγή αφορά τη νέα αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Κατά τους προσεχείς μήνες το Συμβούλιο θα εξετάσει δύο θεμελιώδεις τρόπους για την ενσωμάτωση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη σφαίρα την κοινοτική. Το πρώτο, ε, ο πρώτος τρόπος αφορά το σχέδιο κανονισμού ε, για τη μέθοδο μετάβασης των υφιστάμενων ε, διμερών συμφωνιών και ο δεύτερος είναι η ανακοίνωση της Κομισιόν για τη μελλοντική πολιτική στον τομέα αυτό. Ήδη έχουμε λάβει τι προτάσει τη Κομισιόν στο Συμβούλιο. Μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενημερωθεί για την πρόταση κανονισμού και η Προεδρία μαζί με την Κομισιόν θα φροντίσει να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τι συζητήσει που θα ξεκινήσουν στο Συμβούλιο. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τι συζητήσει με τον πλέον επικοδομητικό τρόπο, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα μείζον ζήτημα και πρέπει να γίνει λοιπόν μια ευρεία συζήτηση και αυτό ίσω απαιτήσει χρόνο. Στόχο μα είναι να κάνουμε την ε, περισσότερη δουλειά επιτόπου και να δώσουμε τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να καταλήξει στι γενικέ ιδέε το συντομότερο δυνατό. Όπω σας είπα και στην αρχή θα ασχοληθώ τώρα και με τις εμπορικές μα σχέσει, με τους βασικούς εταίρους, του κύριου εταίρους. Και μπορώ να πω πολλά πράγματα. Θα είναι βέβαια αυτά αντικείμενο των συζητήσεών μα κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δεν σας εκπλήσει βέβαια το ότι εδώ αναφέρω τι διατρατικέ μα σχέσει τη Ρωσία και την Κίνα. Σίγουρα οι εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες έχουν πρώτη στη σημασία. Το 2009, παρά την δημοσιονομική τη χρηματοπιστωτική κρίση, η Ευρώπη εξήγαγε πάνω από 204 δις ευρώ σε αγαθά, έναντι 159,8 δις εισαγωγών. Στον τομέα των υπηρεσιών, σχεδόν 120 δις εξαγωγές έχουν καταγραφεί σε σύγκριση με 127 δις εισαγωγές. Επομένως, ό,τι αφορά τις άμεσες επενδύσεις, Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολα τα στοιχεία και δείχνουν την αξία και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών μας ε, που καλύπτει μια τεράστια αγορά άνω των 700 εκατομμυρίων ατόμων. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας θα ε, εντείνουμε τις προσπάθειές μας όχι μόνο για να ενδυναμώσουμε την στρατηγική εταιρική σχέση για τα πολυμερή θέματα και για την υλοποίηση του προγράμματος του 2007 για την οικονομική συνεργασία και το ρυθμιστικό διάλογο αλλά και για να αναπτύξουμε έτσι περαιτέρω το έργο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου. Σίγουρα οι σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ είναι καλές. Στόχος μου δεν είναι να μειώσω ή να υποβαθμίσω τα εμπόδια ε, που μας χωρίζουν στον τομέα του εμπορίου. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε για να τα επιλύσουμε. Και θέλω απλά να σας υπενθυμίσω το ότι 98% του εμπορίου λαμβάνει η χώρα χωρίς κανένα πρόβλημα τη χώρα αυτή. Και επίσης ε, όσο πιο ενωμένοι, όσο με, περισσότερο με μια φωνή μιλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο καλύτερα θα μπορούμε να προασπίζουμε τα συμφέροντά μας και τις απόψεις μας. Όπως είναι προφανές ό,τι αφορά τη Ρωσία. Και η Ρωσία είναι στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας μας. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εμπορική σχέση με το σημαντικό αυτό εταίρο και μέχρι πρόσφατα ήταν ε, ανωδική η πορεία του, των εμπορικών μας σχέσεων. Δυστυχώς όμως διακόπη αυτή η τάση λόγω της κρίσης και των μονομερών ε, μέτρων που υιοθέτησε η Ρωσία και τα οποία επηρέασαν το διμερές μας εμπόριο οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στον ΠΟΕ καθώς και διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία που θα αντικαταστήσει την ισχύουσα εταιρική σχέση και συνεργασία και τη σχετική συμφωνία είναι στο επίκεντρο των σχέσεων μας με τη Ρωσία αυτή την εποχή. Όπως φαντάζεστε και εσείς, το Συμβούλιο υποστηρίζει στεναρά την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ και χαιρετίζει τη νέα πολιτική όθηση που έχει λάβει ε, το θέμα αυτό στη Ρωσία. Βέβαια το ε, μπαλάκι είναι ε, στο γήπεδο της Ρωσίας αυτή τη στιγμή και είμαι πεπισμένη ότι αν υπάρξει ε, αν υπάρξουν διατάξεις σημαντικές για το εμπόριο και για τις επενδύσεις, όλα αυτά σε συνδυασμό με την, ε, την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα βελτιώσουν ε, την ε, ποιότητα των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και θα ενταχθούν βέβαια στην εταιρική σχέση για τον εξυγχρονισμό που συμφωνήθηκε στην τελευταία διάσκεψη κορυφής με τη Ρωσία. Βέβαια, σίγουρα το Συμβούλιο υποστηρίζει ταυτόχρονα τη συνέχιση τη δεσμευση τη Ρωσίας για να υπάρξει εξάλληψη των εμποδίων στο εμπόριο, να μην υπάρχουν πλέον τα προστατευτικά μέτρα. Δεν έχουμε τίποτα κατά της Τελωνιακής Ένωσης Ρωσίας, Λευκορωσίας, Καζακστάν. Απλά ε, υπήρξαν κάποιες αρνητικές ε, εξελίξεις και ενδεχομένως να επηρεάσουν αυτός, αυτός ο κοινός δασμός που έχει υιοθετηθεί, ενδέχεται να επηρεάσει τη διαδικασία της προσχώρησης Ρωσίας στον ΠΟΕ και τις διμερείς μας σχέσεις. Έρχομαι στην Κίνα. Είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος μας μετά τις ΗΠΑ σημαντική πηγή, κύρια πηγή των εισαγωγών μας. Και είμαστε και ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κίνας. Η ανοιχτή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε τα μάλα ε, στην ανάπτυξη της Κίνας που βασίζεται στις εξαγωγές. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της ωφελήθηκε από την ανάπτυξη της κινέζικης αγοράς ε, και είναι επιδεκτική ε, σε ένα περαιτέρω άνοιγμα των εμπορικών σχέσεων. Ωστόσο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και η Κίνα εμπορεύεται με δίκαιο τρόπο μαζί μας και ότι σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι τήρησε τι υποχρεώσει στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Σίγουρα ο ανταγωνισμό είναι σκληρό, αυτό είναι γνωστό, είναι σύνηθε, αλλά θα πρέπει να συνάδει και με την ανάγκη να υπάρχει ένα περιβάλλον ε, που δεν θα ευνοεί τι διακρίσει στην κινέζικη αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρει συχνά τι ανησυχίε τη στο πλαίσιο των διμερών επαφών με την Κίνα καθώ και στο πλαίσιο του ΠΟΕ και είμαστε πεπισμένοι ότι συνεχεί διαπραγματεύσεις με την Κίνα για μια ευρεία συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο και στέρεο πλαίσιο για τις διμερεί μας σχέσεις. Ας συζητήσουμε τώρα κάτι στο πλαίσιο του πέμπτου ζητήματος που θέλω να σας αναφέρω, κάτι το οποίο είναι στο επίκεντρο της Βελγικής Προεδρίας. Πρόκειται για την αναπτυξιακή διάσταση του εμπορίου Στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, εγώ θεωρώ τρία είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για την αναπτυξιακή διάσταση πάντα του εμπορίου. Πρώτον, είναι το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων. Δεύτερον, είναι η Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση και τρίτον είναι η Συμφωνία για τι Μπανάνε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, οικονομικέ. Ε, μάλλον ε, συμφωνίε Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, EPAs, με τις χώρες ΑΚΕ. Ο στόχος μας ο βασικός είναι ο ίδιος, δηλαδή πρέπει να συνάπτουμε συνεκτικές περιφερειακές τέτοιες συμφωνίες, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ε, οδηγήσουμε σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και να αναζωογονήσουμε τις εμπορικές ροές από και μεταξύ των χωρών ΑΚΕ. Ιδίω εν ώψη τη παγκόσμια χρηματοπιστωτική οικονομική κρίση που έχει πλήξει τι οικονομίε των χωρών ΑΚΕ και το εμπόριό του. Τώρα, ο ρόλο του Γενικευμένου Συστήματο Προτιμήσεων ε, στο πλαίσιο τη συνολική προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριο και την ανάπτυξη είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σωστά, στο ψήφισμα του Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε το θετικό ρόλο του μέσου αυτού υπέρ και προ όφελο των αναπτυσσόμενων χωρών. Ωστόσο, τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τέλειο και κανείς μπορεί να ε, διαρωτάται, μπορεί να βελτιωθεί το τρέχον σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει αναθεώρηση και πανεξέταση του συστήματος για τους επόμενους μήνες. Συμφωνούμε με την έκκληση του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να τεθεί ε, σύντομα σε ισχύ αυτό το νέο ε, καθεστώς. Είμαστε όμως ως Συμβούλιο και ανοιχτοί στο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο παράτασης Τη ισχύω ε, του τρέχοντος κανονισμού για περιορισμένη διάρκεια για να μην υπάρξει νομικό κενό μέχρι ότου εντριθεί ένα νέο γενικό κανονισμό. Και έρχομαι στη Συμφωνία για τι Μπανάνε, η οποία υπεγράφει πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τι ε, χώρε Λατινική Αμερική αφενός και με τις ΗΠΑ αφετέρου. Αυτή η συμφωνία δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανή τελικά να επιλύσει με επικοδομητικό τρόπο εμπορικέ διαφορέ και δει μια αρκετά μακροχρόνια εμπορική διαφορά. Επίση δείχνει ε, ότι έχει βγει από τη μέση και ένα από τα εμπόδια τα οποία θα πρέπει να επιλύσουν οι διαπραγματευτέ για την ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα. Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για τη συνολική συμφωνία που επετέχθη στη Γενέβη, ότι δηλαδή η συμφωνία αφορά επίσης και αντιμετωπίζει τις θεμητές ανησυχίες των λατινοαμερικανικών χωρών και των χωρών ΑΚΕ ε, για τα τροπικά προϊόντα ε, και το λεγόμενο preference erosion. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα συνοδευτικά μέτρα ε, για τις μπανάνες. Ολοκληρώνοντας ε, με την ατζέντα της Προεδρίας μας, τα πολύ λίγα λόγια για την άκτα, τη συμφωνία ε, την εμπορική συμφωνία για την αντιμετώπιση τη ε, παραποίηση και των απομιμήσεων. Ήδη έχετε συζητήσει το φάκελο αυτό στην Επιτροπή σα δεν θέλω να σας κάνω ιστορική αναδρομή, απλά να τονίσω ότι η αποτελεσματική προστασία των ε, δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία είναι προτεραιότητα η οποία επανειλημμένως ε, έχει αναφερθεί από τα δύο θεσμικά όργανα στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προστασία, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ανταποκρινόμενη ε, στα αιτήματα του Κοινοβουλίου και με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια, ω Συμβούλιο αναλάβαμε έναν προβλεπτικό ρόλο σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του ενοποιημένου σχεδίου του κειμένου ώστε να ενημερωθεί κοινωνία των πολιτών, να ενημερωθούν και οι ενδιαφερόμενοι φορείς για το τι είναι επιτάπητος και το τι δεν είναι επιτάπητος. Το Συμβούλιο χαίρεται που οι, οι άλλοι ε, εταίροι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποφάσισαν επίσης να ανταλλάξουμε απόψεις και έτσι απελευθερώ και κοινά ε, από κοινού μάλλον αυτό το κείμενο. Ένα γύρος διαπραγματεύσεων έγινε στη Λουκέρνη από τις 28 Ιουνίου στην 1η Ιουλίου η έκβαση του γύρου αυτού ήταν ε, ότι οι συμμετέχοντες υπενθύμησαν το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ε, τις πτυχές που δεν καλύπτονται όπως ε, ο κανόνας Three Strikes Rule, το γεγονός ότι η άκτα δεν πρόκειται να, συνάψει νέα, να περιλάβει νέα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή να μειώσει υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Επίτροπος θα μιλήσει σήμερα για την άκτα από ό,τι μου λένε. Βέβαια η άκτα δεν θα παρεμποδίσει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, θα συνάδει με τη Συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ και τη δήλωση για το TRIPS και τη δημόσια υγεία και τέλος δεν θα παρεμποδίσει τη διασυνοριακή διέλευση των θεμητών γενώσιμων φαρμάκων. Ολοκληρώνοντας, θέλω να υπενθυμίσω τη μεγάλη σημασία που το Συμβούλιο ε, προσδίδει στο νέο ρόλο της Επιτροπής σας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας και είμαι πεπισμένος ότι θα έχετε επικοδομητική συνεισφορά η οποία θα οδηγήσει στην επίτευξη ε, του κοινού μας στόχου για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Ολοκληρώνοντα, η κοινή εμπορική πολιτική είναι σε ένα σταυροδρόμι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, έχουμε ένα νέο κεφάλαιο μπροστά μα και το κοινοβούλιο σα, το κοινοβούλιο μα, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η Βελγική Προεδρία θέλει να συνεργαστεί μαζί σα ώστε να επιτελέσουμε τι σημαντικέ αυτέ αλλαγέ που χρειάζονται. Και μαζί στι 31 του Δεκέμβρη θέλουμε, ατενίζοντα προ τα πίσω, να πούμε ότι ναι, είμαστε στο σωστό δρόμο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την μακρά και εντυπωσιακή αυτή παρουσίασή σας των προτεραιοτήτων της Βελγικής Προεδρίας στον τομέα του εμπορίου. Πληροφοριακά, χθες έγινε briefing, ενημέρωση, σχετικά με τον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων άκτα. Ο αρμόδιος επίτροπος ε, βρίσκεται σήμερα εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ όμως, αλλά έχετε δίκιο πράγματι χθες ε, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με την άκτα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στις ερωτήσεις. Επτά ομιλητές έχω στον κατάλογο. Από όλες τις ομάδες από όλες τις πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να περιορίσουμε τον ε, χρόνο παρέμβασης τέσσερα λεπτά το πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκπρόσωπο του ΕΛΚ, την κυρία Κουίστα Ρόβολ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, που ήρθατε εδώ. Ενδεχομένως έχετε πολλά άλλα να κάνετε στις Βρυξέλλες από το να έρθετε εδώ στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είναι πολύ καλό. Υπάρχει αυτή η πολιτική η εμπορική. Κάθε προεδρία ε, περίπου μας λέει το ίδιο πρόβλημα. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Η Προεδρία της Ισπανίας έκανε κάποια πρόοδο, κυρίως με τη Λατινική Αμερική, αλλά έμεινε πίσω σε πολλά άλλα θέματα. Δύο ερωτήσεις, λοιπόν. Εμείς κάνουμε διμερείς διαπραγματεύσεις για να πετύχουμε συμφωνίες. Απ' την άλλη. Λέμε. Δεν εννοείται. Μάλλον άλλη ερώτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας πώς θα μπορούσε να παρουσιάσει κάτι ώστε να προχωρήσει ο γύρος της Δόχα. Από τις περασμένες διαπραγματεύσεις δεν βλέπω κάτι τέτοιο να είναι δυνατό, αλλά ίσως εσείς βλέπετε να υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δεύτερη ερώτηση. Πολύ σωστά είπατε ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αλλάξει ε, τελείως μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και ε, αλλά και εσείς όπως Επίτροπος Δεφίφτε έχετε ήσασταν εξίσου ασαφείς. Εσείς πώς βλέπετε τη συγκεκριμένη συνεργασία και τελευταία παρατήρηση, μάλλον παρατήρηση, με τελευταία παρατήρηση η έκθεση για τις ε, σχέσεις με τη Ρωσία την οποία συνέγραψα όπου διαπιστώνεται ε, ότι η έκθεση αυτή ακόμα ισχύει διότι πολύ λίγα ε, έχουν αλλάξει. Πιστεύετε εσείς ποτέ ότι η Ρωσία θα θέλει να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κατεραρίφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Προεδρία του Βελγίου για την παρέμβαση εδώ. Ε, υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να πούμε. Πρώτα, είπατε με πολύ συγκεκριμένα για τις μερίες συμφωνίες, αλλά η ομάδα μας ε, θεωρεί ότι αυτή η, η πολιτική δεν οδηγεί πουθενά έχουμε μια πραγματικότητα στο παγκόσμιο σύστημα, βλέπουμε δεν λειτουργεί, το Συμβούλιο και οι Επιτροπή συνεχίζουν να συνεχίζουν με το σύστημα των διμερών συμφωνιών που δεν οδηγεί πουθενά. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι η συνεκτικότητα, η συνέπεια των πολιτικών. Πολύ καιρό τώρα υπάρχει μια, ε, ε, μια εικόνα για την πολιτική την εμπορίου η οποία δεν λαμβάνει περίπου καθόλου υπόψη τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν στην έρευνα, στη βιομηχανική πολιτική. Πολιτική εμπορίου θα πρέπει να έχει να κάνει σχέση πάντοτε με, το σύνολο των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Τις επιπτώσεις και την ε, ε, διαδραστικότητα θα λέγαμε τις άλλες πολιτικές. Το βλέπουμε αυτό στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επίσης, ε, στον Επίτροπο Ντεγκίστ ανέφερα ότι, ότι έχουμε το θέμα της ερεύνης. Για παράδειγμα η προσπάθεια να βρεθούν νέους τομείς για την άπτυξη του εμπορίου. Ε, η πρόοδος είναι πολύ περιορισμένη Βλέπουμε δηλαδή ενώ υπάρχουν περιορισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επενδύσει στην έρευνα. Και μήπω θα έπρεπε να, να μας πείτε αν έχετε κάποιο προβληματισμό πάνω σε αυτό το θέμα. Επίση, κάτι ακόμα. Η ομάδα μα θα ήθελε σε όλε τι πολιτικέ, τα διμερείς συμφωνίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια. Θα το δούμε τι επόμενε εβδομάδε. Κριτήρια διαφορετική φύσεως αλλά φυσικά θέματα που αφορούν στην κοινωνική πτυχή, στην περιβάλλον, κριτήρια τα οποία επίσης έχει θεσπίσει ίσως Φιερνής ε, Οργανισμός Εργασίας. Ας μην μπω τώρα σήμερα στις λεπτομέρειες, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτά τα θέματα. Χαίρομαι για αυτά που λέτε όμως Ε, ότι, ότι λέτε ότι δίνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή κάνει μια προσπάθεια, δίνει έμφαση στα συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά εδώ μας παίζεται ένα ντουζ το οποίο θα λέγαμε είναι κρύο ζεστό. Τι λέτε εσείς, σαν Προεδρία του Βελγίου, Εσεί ε, θεωρείτε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι ούτω ώστε να βοηθήσετε φέρει πίνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει περισσότερο σε ορισμένε διαδικασίες πιο επικοδομητικά. Και τώρα για το άκτα και κλείνω. Χαίρομαι για αυτά που είπατε, αλλά έγινε μια ανεπίσημη συνάντηση χθε και έχω ακούσει κάποια πράγματα ε, δεν ήμουν παρόν. Αλλά ήθελα να πω ότι σε τι χρησιμεύει το κοινοβούλιο αν γίνονται συναντήσει και κλειμένο το θηρόν και δεν μπορεί να συμμετάσχει. Αυτό θα ήθελα επίση να μου το πείτε πάνω σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την άκτα δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κάτερα, λέει ο Πρόεδρο. Με την Κάζακ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαιρετίζω και τον κύριο Υπουργό, τον συγχαίρω για την εδώ παρουσία του και την παρουσίαση που έκανε του της ε, Βελικής Προεδρίας. Σίγουρα έχετε φιλοδοξίες να συνεχίσετε ένα θέμα, ένα τομέα ε, στο οποίο έχει κάνει αρκετά η Ισπανική Προεδρία και να υπάρχει συνέχεια. Καταρχήν εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ στους προλαλήσαντες ε, συναδέλφους σοσιαλιστές και ΕΛΚ όσον αφορά για τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Βελική Προεδρία όσον αφορά αυτό τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις νέες αρμοδιότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τα πέτυχε στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνος για τη συνεργασία της Επιτροπής και του Συμβουλίου για να για να, υπάρξει εφαρμογή αυτών των νέων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε, Υπουργό, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ ότι υπάρχουν δυσκολίες στη χώρα σας ε, και είσαστε στην Προεδρία αυτή τη στιγμή, αλλά απ' την άλλη, ίσω ε, ίσως το καθήκον σας να διευκολυθεί από το γεγονός ότι ο αρμόδιος επίτροπος για το διεθνές εμπόριο είναι συμπατριώτης σας. <laughs> Τέλος πάντων. Ο πρόεδρος λέει ότι δεν εκπροσωπεί τις χώρες μέλη. Ε, ε, ε, ο μιλτής λέει το θεωρώ σαν μια τρόπο ανθρώπινης επαφής για τη συνεργασία. Είναι σημαντικό για τις πολιτικές ομάδες να ξέρει κανείς ότι η Επιτροπή στα πλαίσια της συνεργασίας με τις χώρες Mercosur θα συνεχίσει την εντολή της παρόλο που υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις σε ορισμένε χώρες όσον αφορά την εντολή που υπάρχει για τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες Μερκοσύρ, συγκεκριμένα για την ε, ε, Γεωργία. Τι σκοπεύετε να κάνετε, ε, πώς θα το δείτε αυτό στα πλαίσια τη, με την Επιτροπή. Και επίσης να πω για τη ρήτρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές ε, συμφωνίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ορισμένες τρίτες χώρες. Τι γίνεται εσείς προβλέπετε κάτι, θα ενοποιήσετε τις προϋποθέσεις για το πώς ακριβώς δηλαδή, για το πώς θα εφαρμόζονται οι ρήτρε αυτές που έχουν να αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες με τρίτες χώρες, Φερρυπίν με τη Σιριλάνκα. Ευχαριστώ. Ο τους πράσινους τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό. Αν οι πηγές μου είναι σωστές, όταν παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Προεδρίας, αναφέρατε σαφέστατα, δεν θέλετε μια θεατρική, έτσι, ε, εντυπωσιακή πολιτική με 20 φιλοδόξες ε, προσπάθειες, 30 στόχους. Καταλαβαίνω όμως ότι έχετε ένα ευρύ όραμα όσον αφορά την Προεδρία σας και αυτό φυσικά καθορίζει κάποιες προτεραιότητες. Όσον αφορά τη συμφωνία ανάμεσα ε, στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό θυμίο στο οποίο η ομάδα μου θα ήθελε να έχει την γνώμη της Βελικής Προεδρίας. Το θέμα έχει να κάνει με τη συμμετοχή των ε, βουλευτών, ευρωβουλευτών, στις, επιτροπές, σε συναντήσεις συντονιστών σε επίπεδο διεθνών διαπραγματεύσεων. Τι λέτε, η δεν θέλουμε να είμαστε ε, διαπραγματευτές, αλλά ε, παράγοντες οι οποίοι ακολουθούν εκ του συστάδιν τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερο θέμα. Η εταιρική σχέση με το ΣΑΝ. Ξέρετε, μια περίπλοκη, δύσκολη διαπραγματεύση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές τις επιφυλάξεις του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ιδέα να υπάρξει μια συμφωνία ενισιμένη ένα χρόνο μετά την υπατογραφή της εταιρική σχέσης και ανησυχούμε διότι αυτή ε, de facto νέα διαπραγματεύση ε, περνάει τη στιγμή που η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε την άποψή σας όσον αφορά την Βελγική Προεδρία. Θα συνεχίσει με αυτές τις διαπραγματεύσεις με το Τουρκμενιστάν ή όχι. Επίσης αναφέρθηκε το ΑΚΤΑ. Δύσκολη συζήτηση. Και εγώ θεώρησα ότι ε, όταν υπάρχει ένα εμπιστευτικό σύστημα όσον αφορά τα έγγραφα για να μπορώ να ενημερώνουμε εντάξει το καταλαβαίνω αλλά αν θέλει κανείς να κάνει μια δράση πολιτική όσον αφορά το άκτα, ε, ε, είναι δύσκολα. Σε μια συνεδρίαση μπορεί κανεί ίσως να εκφραστεί, αλλά υπάρχει το θέμα του εμπιστευτικού, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε σαν ευρωβουλευτές από εκεί και πέρα. Εσείς τι λέτε από την πλευρά της δημοκρατίας ε, σαν θεσμικό όργανο ευρωπαϊκό. Επίση, αναφέρατε την πολυμερή ε, συμφωνία Περού-Κολομβία. Εγώ θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα συμμετάσχει πριν από το τρίτο εξάμεινο του 2011 δηλαδή. Τι, πώς το βλέπει η Βελική Προεδρία. Μήπως γίνονται γρήγορα αυτές οι διαπραγματεύσεις για αυτή τη συμφωνία. Σε αυτή την Επιτροπή Ξέρετε, έχουμε πολλέ φορέ συζητήσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κοινωνικά δικαιώματα όσον αφορά αυτή τη χώρα. Εσείς, σε σχέση με αυτή την ατζέντα, ε, μήπω θεωρείτε ότι οι διαπραγματεύσει προχωρούν πολύ γρήγορα. Τώρα, στι προτεραιότητε ε, υπάρχει και το θέμα του, του κλίματος, υπάρχει το θέμα του διοξιδίου του άνθρωπος, το θέμα της τεχνολογίας. Όταν δηλαδή συζητάμε για αυτά τα θέματα και υπάρχει και η κλιματική διάσταση, θεωρείτε ότι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό το θέμα όταν έχουμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, κλιματολογικές αλλαγές. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Χέρμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την δουλειά ακριβίας που έχει κάνει. Είχα ήδη σήμερα ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή ε, συνταγματικών θεμάτων και ακούσαμε μια ακριβή περιγραφή των στόχων και του προγράμματος της Βελγικής Προεδρίας ε, με στόχο την επίλυση διαφορών θεμάτων. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι η Βέλγικη Προεδρία έχει προετοιμαστεί πολύ καλά για το εξάμεινο αυτό. Θα ήθελα να τονίσω δύο ή τρία πράγματα, χωρίς να επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν. Θα με ενδιέφερε αν παίρνετε στα σοβαρά τις προσδοκίες του κοινού η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σχέση ε, Συμβουλίου, ε, Κοινοβουλίου και Κομισιόν θα πρέπει να είναι πιο διαφανής και πιο κατανοητή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Τι πιστεύετε όσον αφορά την εφαρμογή των πράξεων εξουσιοδότηση, των διαδικασιών ε, συναπόφασης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της εμπορικής πολιτικής. Συγκεκριμένα μιλάω για τα άρθρα 270-271. Ε, Πολύ συγκεκριμένα, πώς μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Ελπίζω η Βελγική Προεδρία να μπορεί να κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά Λαμβάνοντα υπόψη σοβαρά τι προσδοκίε των πολιτών μα, διότι αυτού δεν τους νοιάζει το ένα ή το άλλο άρθρο. Θέλουν επίλυση των προβλημάτων. Και εάν δεν τα επιλύσουμε αυτά, θα συμβάλλουμε σε μια ε, συνεχή μόνιμη αντίσταση στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενδιαφέρουν ε, λοιπόν οι σχέσεις ε, Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών επειδή είναι οι πιο βασικές ε, δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Επίσης όσον αφορά το θέμα της άκτα, να αναφέρω μία πτυχή. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο οι διαπραγματεύσεις άκτα να πάνε στο πολυμερές επίπεδο, για παράδειγμα στη WIPO ή στον ΠΟΕ διότι το θέμα άκτα επηρεάζει την πραγματικότητα της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες. Τρίτη ερώτηση, να μην μακρηγορήσω. Μίλησατε για τις μπανάνες. Πιστεύετε ότι όταν ε, η ε, ε, Επιτροπή κάνει νέες παραχωρήσεις ε, στην, στο Περού, την Κολομβία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. εγώ είχα ασχοληθεί με το θέμα αυτό ως προς τις χώρες ΑΚΕ. Οι χώρες ΑΚΕ λοιπόν θα έρθουν και θα πούνε τι και με θα γίνει. Η Βελγική Προεδρία συνειδητοποιεί ότι υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση και θα καλέσει την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα των ε, εξαγωγών μπανάνας. Και επίσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο συνάδελφος Ζαντό αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και θα ήθελα να επανέλθω στην πραγματικότητα που ε, κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Κολομβία. Το Φλαμαδικό Κοινοβούλιο απέρριψε συμφωνίες συνεργασίας ε, ιδιαίτερα λόγω των ε, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει νέα προσέγγιση του Συμβουλίου από πλευράς του Συμβουλίου για να επηρεάσει την κατάσταση. οι πολιτικές αυτές πτυχές επηρεάζουν ε, και την, ε, τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες περιοχές του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο William Bartmouth από τους ε, Ελεύθερους Ευρωπαίους Δημοκράτες. Εκτός μικροφώνου, κύριε Ε, ζήτω συγγνώμη. Αναφέρατε την Κίνα. Όταν ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες το φθινόπωρο, ένας καθηγητής του Χάρβαρτ μου είπε ότι στην Κίνα έχουν ανάπτυξη 10%. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε 10% ανεργία για πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες, για πολλές χώρες του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το νούμερο αυτό βρίσκεται πιο κοντά στο 20%. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, να ζητήσω τη γνώμη σας σχετικά με την η τιμή του κινέζικου συναλλάγματος. Ε, πιστεύετε ότι είναι υποτιμημένο? Μήπως θα πρέπει να υπάρξει ανατίμηση του κινέζικου συναλλάγματος. Μήπως ε, η Κίνα ε, ασκεί την πρακτική του μερκαντιλισμού και έχω μια σειρά άλλων ερωτήσεων που θα ήθελα να σας θέσω σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σαν συνέπεια τη συνθήκη τη Λισαβόνα, έχουμε τώρα μόνιμο πρόεδρο του Συμβουλίου, έχουμε επίσης ε, μόνιμο υψηλό εκπρόσωπο. Η ύπαρξη αυτών των δύο θέσεων επηρεάζει τις ε, προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας στον τομέα της διεθνούς εμπορικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη, έχοντας κατά νου ότι η Βελγική Προεδρία θα διαρκέσει μόνο 6 μήνες. Και τέλος, αναφέρατε το GSP+, το GSP -SYN, το Σύστημα Κοινωνικών Προτιμήσεων -SYN, ε, το οποίο θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμένα και κάποιους άλλους συναδέλφους. Μιλήσατε για κάποιες τροποποιήσεις ε, στο σύστημα αυτό. μπορείτε να μας πείτε ποιες θα είναι οι τροποποιήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ε, η συνάδελφος Μουσκαρτίνη, που βρίσκεται στα δεξιά μου, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Ευχαριστώ την πολύ σωστή παρουσίαση του κυρίου Υπουργού. Εγώ θα περιοριστώ σε κάποιες ε, μικρές ε, ερωτήσεις. Είναι δυνατόν η Προεδρία του Βελγίου να λάβει υπόψη το θέμα του εναρμονισμού όσον αφορά τον έλεγχο στα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ όπου ο αγώνας που γίνεται κατά της, παραπημένων προϊόντων και του παράνομου εμπορίου ε, παρουσιάζει όχι μόνο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, αλλά, αλλά ε, ε, ένα γενικότερο πρόβλημα για την επαναλειτουργία, θα λέγαμε, επανασυντονίση της οικονομίας μας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε, η Προεδρία σας θα προσπαθήσει να συντονίσει ένα σύστημα ελέγχου που θα αναμονήσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται όταν έχουμε την, ε, ε, τέτοια προϊόντα που καταλήγουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει, ξέρετε, ε, ένα σύστημα στο οποίο, για το οποίο δουλεύω εγώ για, το, για τον τρόπο ελέγχου ε, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η δράση της ε, Βελικής Προεδρίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εξετάζουμε πολύ προσεκτικά, εδώ και καιρό θα έλεγα, ε, και ε, από το 2005 και μετά η Επιτροπή και αυτή είναι πολύ ενεργή. Προσπαθεί να βρει έναν ορισμό. Μια άλλη πτυχή. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μας ότι η Αφρική ήδη, εδώ και καιρό θα έλεγα, είναι μια ήπειρος η οποία, στην οποία μάλλον η Ινδία και η Κίνα ε, δρούνε πολύ θα λέγαμε επιθετικά που μπορούν να αποσταθεροποιήσουν ε, γενικότερα ε, την κατάσταση. Οι, οι αγορές αυτών των χωρών ε, δημιουργούν ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων στα πλαίσια του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα ένα παράδειγμα όπου βλέπουμε μια, ε, θα λέγαμε μια, ένα θέμη του ανταγωνισμού. Μετά έχουμε τις Mercosur. Ακολουθούμε τη συμφωνία εκ του συστάδινα. Όλοι μας. Όπως ανέφερε και προηγουμένως ένα συνάδελφος. Εμείς ανησυχούμε, το έχουμε εκφράσει αυτό, όσον αφορά την πτυχή που έχει να κάνει με τη Γεωργία. Το Συμβούλιο ε, στα πλαίσια της Βελικής Προεδρίας θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά αυτές τις πτυχές που δεν δείχνουν να αναλαμβάνουν υπόψη αυτή τη στιγμή και είναι επικίνδυνο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ γύρω στον ερωτήσεων. Δεν θέλω όμως και εγώ να θέσω ένα ερώτημα για το γύρο της Δόχα, διότι από ό,τι φαίνεται μόνο λόγια λέμε, ότι επενδύουμε στην ταχεία ολοκλήρωση των ε, διαπραγματεύσεων του γύρου της Δόχας, χωρίς όμως να κάνουμε τίποτα στην πράξη για να επιτυχθεί αυτός ο στόχος. Τι θα μπορούσαμε και τι θα έπρεπε λοιπόν ε, να κάνουμε για να κινηθούν τα πράγματα. Ή μήπως περιμένουμε να ταράξουν τα νερά ΙΠΑ και να κάνουν μια συμφωνία με Κίνα, Βραζιλία, Ινδία. Συμφωνούμε με την άποψη των ΙΠΑ ότι το πακέτο αυτό είναι σήμερα παράδεκτο οι με των μέτρων του 80 και θα πρέπει Κίνα, Βραζιλία και Ινδία να δώσουν περισσότερα σε σχέση με το πακέτο το... και αυτά που του ζητάει. Πως πρέπει να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία με τους άλλους εταίρους και με αυτήν την συμφωνία να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ή να τους περιμένουμε να... και να τους κοιτάμε μέχρι να καταλήξουν αυτή σε συμφωνία. Είναι λίγο δυσάρεστη, άβολη η κατάσταση αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας τόσο σημαντικός εμπορικός εταίρος να περιμένει και να βλέπει τι κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Έχετε πολλές ερωτήσεις να απαντήσετε. Γι' αυτό ε, θα σας δώσω τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά. Νομίζω αρκετό είναι ο χρόνος για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα ήθελα να πάνω να μιλήσω γερμανικά, καταλαβαίνω γερμανικά, αλλά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 Uh, question going sometimes into detail with the Κάποιες φορές έγιναν και κάποιες συζητήσεις στην Επιτροπή 133, 207 έγινε αυτή η Επιτροπή. TPC. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι δύο πράγματα. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση πρώτα απ' όλα, η συνθήκη της Λισαβόνας είναι πολύ πιο ξεκάθαρη και ρητή και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Και έπειτα υπάρχει στο τέλος η έγκριση που θα πρέπει να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν μπορούμε και να φανταστούμε καν ότι δεν θα ακούμε τη γνώμη του Κοινοβουλίου όταν εκφράζεται αυτή μέσω ενός ψηφίσματος ή μέσω μιας ακρόασης όπως αυτή και ότι οι επίσημες, ανεπίσημες λοιπά επαφές θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν για να έχουμε, πώς να το πω, την σχέση, τη διασύνδεση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Ε, να προσέχουμε τώρα όσον αφορά του διαμαρπαντευτέ να είναι θα λέγαμε ε, συμμετέχοντες ενεργά. Θα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να έχει τη θέση ότι δεν ε, διαπραγματεύεται ότι είναι λίγο περιορισμένη θέση του. Η, θέση του είναι να ελέγχει, να πει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν συμφωνούμε, αλλά, αλλά δεν εντάσσεται συλλογική ότι, ε, ότι είναι διαπραγματευτής. Είναι βασική θέση αυτή, κύριε Πρόεδρε. Η ενημέρωση είναι η βάση όλης της σοφίας. Να υπάρχουν πολλές ανταλλαγές ε, απόψεων και στο τέλος, τέλος πάντων να υπάρχει μια ε, συμφωνία, να υπάρχει σύμφωνη ή όχι γνώμη του Κοινοβουλίου και φυσικά να εφαρμόσουμε αυτό που λέμε best practices. Φυσικά ε, να εισακούεται το Κοινοβούλιο, αλλά να καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Ξέρετε, το κοινο το, το Βέλιο έχει μια παράδοση ε, όπου υπάρχει πάρα πολύ ε, θα λέμε ομοσπονδιακής προσέγγισης, ε, προσέγγιση σε πολλά θέματα και ο καθένας έχει τις, ε, τις ε, αρμοδιότητες του. Σχόλιο τώρα του Προέδρου, εκτός μικροφώνου η ερώτηση, λέει, ε, λέει ότι ναι καταλαβαίνει, είδε το χαμόγελο της κυρίας, αλλά δεν έχουμε ακούσει το σχόλιο της κυρίας. Τέλος πάντων, άκουσα πολλά ενδιαφέροντα σχόλια. Και επίσης λέτε ότι η λογική του υπάρχει μια συνεκτικότητα όσον αφορά τις πολιτικές. Ξέρετε ότι έχουμε την Προεδρία η οποία έχει τις αρμοδιότητες της αλλά υπάρχει και ο πρόεδρος του Συμβουλίου για τις ε, Γενικές Υποθέσεις, ο οποίος έχει και αυτός την αρμοδιότητα να πετύχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συντονισμό στις διάφορες δράσεις. Ε, Όντω, δηλαδή υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να υπάρχει ένα συντονισμό όσον αφορά τι διάφορε ευρωπαϊκέ πολιτικέ, αλλά α μην μπω τώρα σε λεπτομέρειε. Έχετε όμω δίκιο. Όταν λέτε επίση την έμφαση πρέπει να δοθεί στην έρευνα, εγώ το μόνο που έχω να πω ότι είναι σαφές ότι στην Ευρώπη πρέπει να δοθεί μια ε, περαιτέρω έμφαση όσον αυτό το θέμα. Κύριε Καζάκ τώρα. Α, εκεί είσαστε. Κοιτάξτε. Τι, μιλήσατε στα γαλλικά. Α, ναι. Και ξέρετε, αυτό που θα ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι ε, Εμεί δεν είμαστε μια κυβέρνηση, είμαστε μια προεδρία η οποία διαδέχεται μια άλλη και έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν είμαστε πολιτικοί πολιτικοί, καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. το ότι ο πρόεδρος είναι, ε, συγγνώμη, ο επίτροπος αρμόδιος είναι Βέλγος δεν αλλάζει τίποτα, είναι Ευρωπαίο επίτροπο. Να γίνει κατανοητό. Τώρα κάτι άλλο για το Μερκοσύρα, αν δεν Για τη Γεωργία Υπάρχει μία μόνο συνεδρίαση, υπήρξε ένα briefing και δίνουμε έμφαση, τι λέει εδώ στη ρήτρα, τι, α, για τα θέματα της Γεωργίας. Ε, κοιτάω εδώ τα σχόλια που κάνατε και θα λάβουμε υπόψη αυτά που λέτε. Απάντησα σε μια σειρά ερωτήσεων. Τώρα, το Τουρκμενιστάν. Δεν έχω προετοιμαστεί για αυτό το θέμα είχατε την εντύπωση, ακούοντάς σας, για το Τουρκμενιστάν, ότι έχουμε το θέμα πώς μπορεί αυτή η πολιτική εμπορική να χρησιμοποιηθεί, αν κατάλαβα καλά, να αποτελέσει μοχλό για να ασκηθούν κάποιες πιέσεις και για να ενταχθεί στη γενικότερη πολιτική, εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι, αν κατάλαβα καλά, το θέμα για το Τουρκμενιστάν ή να μου ξαναεξηγήσετε το πραγματικό πρόβλημα ή αποδέχεστε αυτό που είπα για το ερώτημα που κάνατε. Ε? Δεν ναι, προετοιμάστηκα σωστά η αλήθεια πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, Κολομβία, Περού. Δεν υπάρχει καθυστέρηση, ούτε επιτάχυνση. Από πού σου. Που δρα αρνητικά. Άλλοι συνάδελφοι αναφέρανε το θέμα της βελικής κυβέρνησης όπου κάποιες περιοχές αποφάσισαν να έχουν μια επιφύλαξη όσον αφορά την Κολομβία. Είναι σημαντικό θέμα, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ε, ενσωματώνουμε τις διάφορες προτεραιότητές μας δύο τινά Πρώτο, δεν θα πρέπει να είμαστε τυφλοί απέναντι στην πραγματικότητα ότι η ύπαρξη του εμπορίου αποτελεί κάτι που επηρεάζει θετικά το κοινωνικό κλίμα καθώς και τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Ή τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζει κανείς το επιχείρημα ότι η μη ύπαρξη εμπορίου δεν είναι απαραίτητο καλύτερη για τις κοινωνικές ε, ε, και άλλες προτεραιότητες που προβάλλουμε. Δεν, δεν θέλω να πιστεύετε ότι αυτή είναι εύκολη ε, απάντηση, αλλά η ύπαρξη εμπορίου με κάποιον εταίρο μπορεί να αποτελεί την ε, αρχή μιας κατάστασης όπου να μπορεί να ζητήσει κανείς κάτι ως αντάλλαγμα. Και επίσης οι συμφωνίες νέας γενιάς περιέχουν ρητές αναφορές στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει αναφέρει αυτό. Συχνά αυτό που λείπει είναι η παρακολούθηση. Η διασφάλιση της ε, συμμόρφωσης με αυτά που συμπεριλαμβάνονται στη, σε μια τέτοια συμφωνία. Η κατάσταση δεν είναι πάντα τέλεια. Χρειάζεται βελτίωση. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε τη μόχλευση που θέλουμε στην, στις συζητήσεις ε, τις εμπορικές. Κύριε Σόλς, όσον αφορά τις διοργανικές σχέσεις και τις πράξεις κατεξουσιοδότηση, επιτρέψτε μου. Να σας πω στον χρόνο που έχω. Χθε είχα μια συζήτηση με τον Επίτροπο Σιωφκοβίτς για ακριβώς αυτό το πολύπλοκο θέμα των πράξεων εξουσιοδότηση και της επιτροπολογίας. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με κατάλληλο τρόπο για να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα από τη μία και την διαφάνεια και δημοκρατική νομιμότητα από την άλλη. Δεν είμαι βέβαιος ότι η άκτα σήμερα θα πρέπει να μεταφερθεί στο πολυμερές επίπεδο. Το έχουμε προσπαθήσει και ο λόγος που η άκτα προχωράει με την ταχύτητα που προχωράει δεν είναι επειδή λείπουν περισσότεροι εταίροι. Αν γίνει πολυμερής ε, δεν θα λυθούν απαραίτητα τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Ήδη αναφέρθηκα στην Κολομβία. Κύριε Μπάρτμουθ, με ρωτήσατε για το συνάλλαγμα της Κίνας. Θέλω να ε, παίξω το ρόλο μου σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και νομίζω ότι κάποιες από τις ερωτήσεις που θέσατε ε, δεν ε, είναι θέματα, κάποιες από τις ερωτήσεις που θέσατε δεν είναι θέμα που θα πρέπει να απαντήσει η, ε, η προσωρινή Προεδρία. Η ισοτιμία του κινέζικου με τα άλλα συναλλάγματα σήμερα επηρεάζει την ε, ανάπτυξη που γνωρίζει η Κίνα, η οποία κινείται με βάση τις εξαγωγές. Ταυτόχρονα, έχει ανακοινώσει η Κίνα και έχει στείλει σαφή μηνύματα ότι θέλει να αποκαταστήσει μια κάποια ισορροπία στον κόσμο. Αυτό ωστόσο θα πρέπει να γίνει με αργό τρόπο και όχι με δραστικό. Πολύ σωστό είναι αυτό, αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι ανισορροπίες αυτές δεν θα αλλάξουν από εν μία νυχτή. Με ρωτήσατε επίσης σχετικά με το ρόλο του Χέρμαν Φαν Ρόμπεϊ και της Κάθριν Άστον. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε με την παρατήρηση αυτή. Ε, μου δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβω κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργό μου, εγώ και όλοι οι Υπουργοί της Βελική κυβέρνηση λέμε εδώ και πολύ καιρό. Θέλουμε η Βελική Προεδρία να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη λογική της συνθήκη της Λισαβόνα. Αυτό δεν αποτελεί έλλειψη φιλοδοξιών για την ε, ε Προεδρία μια τέτοια προεδρία μπορεί να συμβάλλει στη διοργανική συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το, την Κομισιόν και το Συμβούλιο και μεταξύ όλων των νέων φορέων ε, που δημιουργούνται με, την, ε, με τη θέση του μόνιμου Προέδρου και του ε, υπατοπροσώπου. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα αυτά, αλλά η Προεδρία δεν θεωρεί ότι έχει ρόλο ηγεσία. Μάλλον εξυπηρετεί, μάλλον τρέχει από πίσω να φροντίσει να μην καθυστερεί κανείς, να μην μένει κανείς πίσω. Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό τώρα με τη δική μας Προεδρία, διότι θέλουμε να δούμε την εφαρμογή της συνθήκης τη Λισαβόνας και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να το πετύχουμε αυτό και στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής, όπου είναι σαφές ότι κάποιες από τις αλλαγές στις αρμοδιότητες Κοινοβουλίου και Κομισιών έχουν αλλάξει σημαντικά. Τι ξέχασα, το GSP... Ξέχασα κάτι. the, Το Συμβούλιο προσλέπει στην ε, παρουσίαση της ε, Κομισιόν της ε, πλήρους αναθεώρησης του ε, του σχεδίου GSP, του Συστήματος Γενικών ε, Προτιμήσεων. Φυσικά περιμένουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γρήγορη υιοθέτηση, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ολοκληρωτικό ολοκληρωμένο και ε, λειτουργικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ε, ανάγκες των χωρών. Πετάω λοιπόν το μπαλάκι στην Κομισιόν, διότι αυτοί θα υποβάλουν έγγραφο και θα το εξετάσουμε όταν θα είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι κλείνουμε τη συζήτησή μας αυτή. Δεν ε, είχαμε προβλέψει δεύτερο γύρο και δεν έχω το χρόνο να δώσω το λόγο σε άλλους ομιλητές. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο μας, τον ε, Βέλγο Υπουργό, για την παρουσίασή του των προτεραιοτήτων της Βελγικής Προεδρίας. Γνωρίζουμε τώρα καλύτερα τις ε, πολιτικές προτεραιότητες και φυσικά δεν είναι η τελευταία φορά που θα μας επισκεφτεί ο Υπουργός Εμπορίου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to you. You get my letter? Uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πριν λοιπόν από την συνάντηση των συντονιστών πρέπει να τα διεκπαιρεώσουμε. Έχουμε δηλαδή το σημείο 5 και οι δυνατόν και το 7. Ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο 5. να με παρακαλώ θέλω την προσοχή σας. Παρακαλώ, σιωπή. Θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2011. Όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Ξετάζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητού μας Πέτερ Στάσνη από το Ευρωπαϊκό Λεκοκόμμα. Κόμμα η, αποφασί η Επιτροπή μας, όπως ξέρετε, αποφάσισε να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο προπολογισμού 2011. Αρμόδια καθήλων επιτροπή, βέβαια, Επιτροπή Προπολογισμών. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή Πέτερ Στάσιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα Θα ήθελα να σας κάνω μια επισκόπηση της γενικής κατάστασης. Προτείνει συνολικά 142,6 δις σε δεσμεύσεις ανάληψης υποχρεώσεων το αύξηση 0,8% σε σχέση με το 2010. και δεσμένε πληρωμών αύξηση κατά 5,8% γύρω στα 130 δις. Σε σχέση τώρα με το GNP, ένα 14% του ΑΕΠΑ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, 1,04%. Το σημαντικότερο, το 45% δηλαδή, 65,4 δις ε, θα πάνε για, για μέτρα θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξης για να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά αυτό το χαιρετίζει γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττεται από την χρηματοπιστωτική κρίση για το 1β ανάπτυξη απασχόληση συνοχή έχουμε μεγάλη αύξηση πληρωμές συν 16,9%. με βάση την εξήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό σχετίζεται με τις ενδιάμεσες πληρωμές για το 2007 και το, την περίοδο μάλλον 2007-2013 έναντι των πληρωμών 2000, 2000. Σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις στο 3 για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης στον τομέα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αύξηση 12,8% δεσμεύσεις ε, πληρωμών επίσης αυξάνουν το 15,4%. Στο 4 τώρα, η Επιτροπή στην πρότασή της σε ό,τι αφορά τον τίτλο 4 Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος εταίρος 8,6 εκατομμύρια σε ε, υποχρεώσεις ένα μικρό περιθώριο 70 εκατομμύρια 0,9% παραμένει. Υπάρχει αύξηση 16% επίσης ε, MFA. Αλλάζουν βέβαια τα πράγματα. Έγινε συνεδρίαση της Κορεπέρη την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς μόνο το ψήφισμα ε, λάβαμε. Δεν ξέρουμε τα νούμερα. Σήμερα θα τα έχουμε στη διάθεσή μας. Παραμένει το πρόβλημα πάντως που είχαμε. macro financial assistance for structural reforms in countries. Τώρα, προέλευση κονδυλίων για τα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα. Έχουμε 25 εκατομμύρια ευρώ από τα περιθώρια του τίτλου 4 και 13 εκατομμύρια από την ε, μεταφορά στο πρόγραμμα DCI και 5 εκατομμύρια ευρώ θα αναπτυχθούν από το χρηματοδοτικό μέσο της πολιτικής προστασίας που θεωρώ ότι με τα συνοδευτικά αυτά μέτρα οι λιγότερες, οι πιο φτωχές, μη αναπτυγμένες χώρες θα ωφεληθούν. Δεν υπάρχει αλλαγή λοιπόν σε σχέση με τα προηγούμενα που είχε φάσει σκορεπέ. Σε ό,τι αφορά τις προσπαρασκευαστικές ενέργειες υπάρχουν τρία ε, business Center Projects που, χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης. Ένα στο Πεκίνο, ένα με τέσσερις θέσεις, με τέσσερις προπολίσεις, Ινδία, ΑΣΕΑΝ ε, και Trade Center ε, στην Ταϊλάνδη. αυτό, αυτό το Trade Center θα μπορέσει να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα πλήρες υπηρεσίες, της ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει αυτό να εξασφαλιστεί στο μότερο δυνατό. Προτινόμενη νομική βάση τα μέσα ICI. Εγώ πριν από λίγα χρόνια εργαζόμουν ε, για αυτή την πολύ σημαντική επένδυση και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαιτέρως. για αυτή την απόφαση θα έχουμε πολλές εξελίξεις σε εκβιομηχανισμένες χώρες, Ινδία, Κίνα, προβλέπουμε αύξηση της τάξης του 10% και περισσότερο και είναι πολύ σημαντική επένδυση λοιπόν για το μέλλον εκεί, για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και για την απασχόληση. Ο προπολογισμό βέβαια δεν είναι μόνο νούμερα. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα έχει δώσει νέε αρμοδιότητε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να σεβαστούν πλήρω τη νέα κατάσταση. Το Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εφαρμογή και εκτέλεση του προπολογισμού, ιδίω στον τομέα της μακροοικονομική ενίσχυση, των μέσων για τι εκβιομηχανισμένε χώρες, της ε, βοήθεια που σχετίζεται με το εμπόριο και ιδίω ε, τη βοήθεια για το εμπόριο. Σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει ε, μία έκθεση παρακολούθησης για το Aid for Trade ε, για την εκτέλεση του 2008 όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των προηγούμενων διαδικασιών κατάρτισης του προπολογισμού. Το ίδιο ισχύει βέβαια ε, και για το MFA, δηλαδή τη μακροοικονομική βοήθεια, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς δαπανώνται οι πόροι για, τα, για τις πιστώσεις αυτές. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα πλαίσιο, ε, ένας κανονισμός συναπόφασης για τη μακροοικονομική βοήθεια, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία, διαφάνεια και παρακολούθηση. Η πρόταση τροποποίηση του κανονισμού ε, για τη για το μέσο των εκμηχανισμένων χωρών είναι επίσης μια θετική πρόταση και ελπίζουμε να λυθούν τα προβλήματα ώστε να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το μέσο αυτό. Σε ό,τι αφορά μια νέα δράση θα έλεγα ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν τα σαντευτικά μέτρα για τις μπανάνες με προτεραιότητα τις πιο φτωχές, ε, αναπτυγμένες χώρες, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Υπάρχουν κάποιε χώρε που εφαλούνται και δεν είναι πια και σε τόσο δίνη κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τώρα τον προπολογισμό, θα μπορούσα να πω ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν απαραίτητε δεσμεύσει, ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να εκπληρώνει τι υποχρεώσει που απορρέουν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και θα πρέπει να λαμβάνεται ιδίω υπόψη η κοινή εμπορική πολιτική. Επίση, θα πρέπει να μπορούμε να συνεισφέρουμε πλήρω στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ. Εν συντομία, Πρόεδρε, πριν ολοκληρώσω, επειδή έχουμε αυτά τα νούμερα και τις αλλαγές που προέκυψαν σήμερα από τη συνεδρίαση της ΚΟΡΕΠΕ της προηγούμενης εβδομάδας, να πω ότι κατέληξε σε μείωση του προπολογισμού 788 εκατομμύρια ευρώ στις αναλήψεις υποχρεώσεων και 3,6 δις για τις αναλήψεις πληρωμών. Δύο δίσες επιστώσεις πληρωμών προτείνεται να ληφθούν από τον τίτλο 1, βιώσιμη ανάπτυξη, και 600 εκατομμύρια από τον τίτλο 2, φυσική πόρη. Πρόκειται για δραματικές περιστολές στι πιστώσει Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό είναι δικαιολογημένο εφόσον η Ευρώπη πλήττεται από την κρίση σήμερα και ιδίω ό,τι αφορά το τίτλο Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στον τίτλο 4, Ευρωπαϊκή Ένωση Παγκόσμιο Εταίρο, σε προτινόμενε περιστολέ 94 εκατομμύρια ευρώ στι αναλήψει υποχρεώσεων. Υπάρχει και μια μικρή μείωση και στο μέσο ICI. Αλλά για το SCI συν ε, δεν θα έχουμε αλλαγή και η μακροοικονομική βοήθεια, τα είπα και πριν. Προτείνεται μείωση 15% και στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές. Θέλω τέλος να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή ΙΝΤΑ θα γνωμοδοτήσει για το σχέδιο του προπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, όπως αποφασίστηκε στις 16 και 17 Μαρτίου και όχι μόνο για το τμήμα 3 του προπολογισμού που καλύπτει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες ε, στη διαδικασία λόγω της νέας διαδικασία ε, προπολογισμού, που ισχύει από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνας. Draft, ε, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε τη γνωμοδότηση στους φακέλους σας. Θα κηρύξω, ξηρίξω την άξιση της συζήτησης τώρα. Ο κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή θεωρώ δεν, μπορέσα, δεν δουλέψαμε ποτέ σε αυτό το θέμα. Αλλά όπως ξέρετε δεν αλλάζει κανείς την ομάδα που κερδίζει. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, και θυμάμαι ότι είχα καταθέσει μια σειρά προτάσεων, κάποιες νήξεις που εκπροσωπούσαν και την ομάδα των Πρασίνων Χαίρομαι όπως ανέφερε αυτά τα διάφορα θέματα, μπανάνες και τα λοιπά, ο Πέτερ, συνεργασία, εμπόριο και τα αλλά κάποιες διευκρινήσεις να κάνω. Θα ήθελα να πω, ο διάβολος βρίσκεται σε λεπτομέρειες. Είχα συντάξει κάποιες παρατηρήσεις. Δεν αναφέρει για το θέμα της μπανάνας ότι θα χρηματοδοτηθεί, η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ταμείο για την ε, Ανάπτυξη. Επίσης, να ζητηθεί από την Επιτροπή ε, για το θέμα της συμμετοχής του Κοινοβουλίου και εγώ αν θυμάμαι καλή είχα προτείνει ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα για να γίνει σεβαστό το δικαίωμα του Κοινοβουλίου. Επίσης, είναι σημαντικό κατά με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 Υπάρχει άλλος που θέλει το λόγο. ο κύριος Σόλς. Ε, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων αυτή ε, για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, όσον αφορά τον προσανατολισμό της Επιτροπής Προϋπολογισμού για τα θέματα εμπορίου, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο το σημείο 2, διότι δεν είναι πολύ σαφές τι θεωρεί η Κομισιόν σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι θα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πώς μπορούμε να ε, ε, να χρηματοδοτήσουμε αυτό το πρόβλημα, το Aid for Trade για παράδειγμα ή άλλα. Ε, δεν ήταν πολύ σαφές αυτό για μένα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς. Θα πρέπει να ζητήσουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Όσον αφορά το σημείο 7, θα ήθελα να προτείνω να να ζητήσουμε και εδώ διασαφήνιση, διότι αν δεν πούμε με ποια κριτήρια χρηματοδοτούμε όσον αφορά τον ΠΟΕ, δεν θα είναι πολύ σαφές αυτό. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καθορίσει το πολιτικό πλαίσιο που να επιτρέπει σε τέτοιες αντιπροσωπείες να συμμετέχουν στις εργασίες του ΠΟΕ. Μιλώ δηλαδή για τους προσώπους των χωρών ΑΚΕ. Επίσης, είναι απαραίτητο να καλυφθούν έξοδα ταξιδίου για εκπροσώπους ε, τουλάχιστον 30 χωρών ΑΚΕ κοινοβουλευτικών. Έτσι να διευρύνουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις χώρες αυτές στον ΠΟΕ. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε αν εννοούμε στα σοβαρά ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις ε, διαπραγματεύσεις ε, στα πλαίσια του ΠΟΕ να ε, ξεφύγουν από το αδιέξοδο και συγκεκριμένα για τον γύρο διαπραγματεύσεων Δόχα. Ε, από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την πολύ πλήρη παρουσίασή του για το σχέδιο προϋπολογισμού 2011. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στην γενική παρουσίαση. Όπως εξήγησε ο εισηγητής, ε, ο προϋπολογισμός επικεντρώνεται στην οικονομική ανάκαμψη. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα σε επίπεδο της Κομισιόν όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το εμπόριο. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, υπάρχει συνέχεια. Η... Πρόκειται λοιπόν για λίγο πολύ τον ίδιο προϋπολογισμό με πέρσι. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποιες πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις που έγιναν από τους ε, βουλευτές. τα θέματα αυτά συζητώνται και σε άλλες επιτροπές, ιδιαίτερα την Επιτροπή Προϋπολογισμού και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο συνοδευτικό μέτρο για τις μπανάνες. Όσον αφορά τον διορθωτικό προϋπολογισμό 2010, ήδη αυτός εξαρτάται από την πρόταση της Επιτροπής 2011, αλλά σημειώνουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν εδώ προβλέπεται ότι 10 χώρες θα επωφεληθούν από το ε, πρόγραμμα αυτό και νομίζω ότι οι 10 χώρες ΑΚΕ θα είναι επιλέξιμες. Η δεύτερη παρατήρηση που μπορώ να κάνω από πλευρά της Κομισιόν έχει να κάνει με την προπαρασκευαστική δράση Ινδία-Κίνα. Η Κομισιόν πράγματι σχεδιάζει στο μέλλον μετά το 2011 συνεχή χρηματοδότηση στα πλαίσια του ICI+. Ε, πρόκειται για ένα μελλοντικό κανονισμό που δεν έχει εκριθεί ακόμα. Συμμεριζόμαστε τη θέση του εισηγητή ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχής χρηματοδότηση για να διασφαλιστεί η λειτουργία του κέντρου αυτού που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά από πλευρά Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πίτερ Στάσνη, έχετε να κάνετε κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα θα ήθελα να, σας να ευχαριστήσω του συναδέλφου για τις παρατηρήσεις τους, ε, να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλ. Κάποιες παρατηρήσεις ε, χρήζουν διευκρίνησης. Ε, είχαμε συζητήσεις με τον ε, David Μάρτιν στο παρελθόν. Ε, μπορεί να συμφωνούμε κάποια πράγματα με άλλα όχι. Όσον αφορά όμως την προσαρμογή και τα συνοδευτικά μέτρα, όλα αυτά αποτελούν άμεσε συνέπειες των νέων συμφωνιών στα πλαίσια του ΠΟΕ και έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τις στοχές χώρες. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρούμε τα χρήματα ε, συμμετέχω και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και σχεδόν ε, είχαν τρελαθεί για να βρούνε ε, τα επιπλέον εκατομμύρια που χρειάζονται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιήσουμε όλες τις χώρες αυτές. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επενδυθούν σε νέες καλλιέργειες για να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά οι χώρες αυτές. Υπάρχουν άλλες περιοχές που παράγουν μπανάνες οι οποίες όμως είναι σχετικά πλούσιες. Οι συνέπειες για τις περιοχές αυτές λοιπόν ε, θα υπήρχαν εμένα, αλλά δεν θα ήταν τόσο δραστικές όσο για άλλες ε, περιοχές. Ε, όσον αφορά το ICI στον κύριο Σόλς, ε, αυτό ε, έχει υποστεί περικοπές ε, κατά ένα εκατομμύριο, αλλά Όπως και στο παρελθόν υπάρχει πάνω από μισό εκατομμύριο για τις δραστηριότητες αυτές και πάντα αποφασίζει η Επιτροπή μας. Σχετικά με τη χρηματοδότηση για την οποία αγωνιστήκαμε αρκετά χρόνια. Το θέμα αυτό συνδέεται στενά με τις δραστηριότητες του ΠΟΕ, όπου και αν ε, πραγματοποιηθούν η δική μας Επιτροπή πάντα όταν αποφάσιζε πετύχαινε πολύ σωστή ισορροπία. Και φροντίζαμε να έχουμε την εποπτεία στο όνομα των εκλογέων μας. Η όλη διαδικασία λοιπόν τελικά θα υποτίθεται ότι είναι προς όφελος των πολιτών. Μπορείτε να συντομεύσετε ε, την επανεμβασή σας. Μόλις τελείωσα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 5η Αυγούστου φέτος το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές δεν επηρεάζουν το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα. Ας προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 7 εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που την χάνουν δημόσια στήριξη. Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων θα έχουμε. Όσον αφορά τις εξαγωγές αυτές ρυθμίσεις, ε, ο εισηγητής μας, ο Γιάννη Ξεντό από τους Πράσινους, θα παρουσιάσει ένα έγγραφο εργασίας που βρίσκεται στον φάκελό σας. Γιάννη Ξεντό, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, πριν να ξεκινήσω, πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε. 15, λεπτά, το πολύ 20. Είναι ένα θέμα νομοθετικής φύσεως. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι παρόντες. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε σε αυτή τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων να συζητήσουμε ε, πριν να γίνει η μεγάλη συζήτηση. Δεν θα μπω τώρα στο, στις λεπτομέρειες του εργασίας να πω ποιος είναι ο στόχος που ορίζει κανείς σαν εισηγητής. Σήμερα έχουμε υπηρεσίες πιστώσεων στις διάφορες χώρες μέλη που δουλεύουν πάρα πολύ ευρέως σε βάση εθνική και οι οποίες υπηρεσίες μέσα από διαπραγματεύσεις μέσω της Επιτροπής συμμετέχουν σε μια ρύθμιση. Ε, μας οδηγεί σε μια κατάσταση. Ε, και τη στιγμή τώρα μάλιστα που λόγω της ε, ε, συνθήκης της συν είμαστε συνομοθέτες, όπως και στα πλαίσια του ΩΣΑ, καταλήγουμε σε μια κατάσταση, τη στιγμή που έχουμε συζητήσει εδώ και πέντε χρόνια, να ε, αντιμετωπίσουμε καταστάσεις οι οποίες ήδη έχουν αριθμιστεί και έχουμε την εξής δυσκολία, δηλαδή να δούμε πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα το Κοινοβούλιο. Για μας το θέμα ε, έχει να κάνει ότι βρισκόμαστε στα πλαίσια μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης όπου οι χώρες μέλη είναι οι βασικοί οι εταίροι που υποστηρίζουν τις βιομηχανίες και μέσα υπηρεσιών για τις πιστώσεις, για τις ε, εξαγωγές και αυτό γίνεται λοιπόν ε, σε όλη την Ευρώπη. Οπότε το, θέμα είναι σε μια Ευρώπη των 27 χωρών τι ακριβώς έχουμε, τι στοχεύουμε. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε μια ε, διαφάνεια, να ξέρουμε τι γίνεται στα επίπεδα αυτών των υπηρεσιών πιστώσεων. Ήδη έχω συζητήσει και είχα επαφή με τον Σιώδη Συγητή. Έχουμε κάνει τις παρα... κατάλληλες ανταλλαγές απόψεων. Η μεγαλύτερη τέτοια υπηρεσία είναι η Αμερικανική. Αυτό που ζητάει κανείς από εμάς τους Ευρωπαίους στην... Ε, είναι να υπάρξει μια εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να έχουμε μια διαφάνεια. Να ξέρουμε ποια είναι τα ρίσκα, και, και αλλά αυτό που διαπιστώνουμε είναι αυτό που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που γίνεται στην αντίστοιχη υπηρεσία της Αμερικής. Θα θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε ποιες είναι, ε, ποιο είναι το ρίσκο σε διάφορα ε, προγράμματα τα οποία ξεκινάνε, επιπτώσεις ε, οι οικολογές, θέματα που να κάνουν με το πετρέλαιο, και όλες οι συναφείς πτυχίες. Δεν θα επεκταθώ, περιορίζουμε σε αυτό, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που θέλουμε εμείς, τροποποίηση των κριτηρίων, όχι, δηλαδή, συγγνώμη, όχι να ακριβώ αλλάξουμε τα κριτήρια, αλλά να, κάνουμε, να πετύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Μεγαλύτερη ορατότητα. Ευχαριστώ. Κάσπαρη uh, ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις ε, εξηγήσεις του. Η στήριξη των εξαγωγικών πιστώσεων είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πολλά κράτη-μέλη έχουν εισάγει το σύστημα αυτό και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πρόθεσης των εξαγωγών. Αλλά μία θέση του εισηγητή μας ε, δεν τη συμμερίζομαι. Δεν πιστεύω ότι είναι πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι θα ε, οδηγήσει σε περιβαλλοντικά προβλήματα ή ότι θα έχει αρνητικέ συνέπειε ε, στα περιβαλλοντικά πρότυπα το ε, μέσο αυτό, διότι στα κράτη-μέλη έχει εφαρμοστεί πολύ προσεκτικά το μέσο αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή μας ε, τι συζητάμε σήμερα. Νομίζω ότι συζητάμε μία λεπτομέρεια Ε, αλλά τελικά θα ψηφίσουμε την έκθεση στο σύνολό της ε, και σίγουρα μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό, να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας Αλλά μιλάμε, αυτή, αυτή τη στιγμή συζητάμε μια τεχνική λεπτομέρεια, να μην παραφουσκώσουμε λοιπόν ε, το θέμα, να ε, γνωρίζουμε ότι απλά συζητάμε μια τεχνική λεπτομέρεια. Και κάποια άλλη στιγμή να συζητήσουμε επί της αρχής το θέμα των εξαγωγικών πιστώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν συμφωνώ με τον Αστάν. Δεν έχουμε, έχουμε να κάνουμε με μια έκθεση μόνο τεχνικής φύσεως. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας λόγω της συνθήκης για να επέμβουμε στην ουσία σε σχέση με αυτά που μας προτείνουν και στις αποφάσεις που θα λυθούν. Ε, μέσω του συστήματος ε, πιστώσεων για τις εκλογές, οι υπηρεσίες χρηματοδοτούν ε, διάφορα προγράμματα με τις εξορίξεις, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και είναι το διπλάσιο από αυτά που κάνει κανείς σε επίπεδο διμερών ε, συμφωνιών υποστηρίζουν την ανάπτυξη. Θα πρέπει όμως να γίνουν κάποιες αλλαγές που οδηγούν σε μια διαφάνεια και στην διάδοση των δεδομένων. Να δει κανείς πώς γίνεται η επιδότηση αυτών των ε, εξαγωγών. Να δει κανείς αυτές τις συμφωνίες. θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεπερνάμε απλώς πέρα για πέρα την πτυχή που είναι καθαρά τεχνικής φύσεως, αλλά έχουμε να κάνουμε πολιτικής φύσεως ερωτήματα. Υπάρχουν συμφωνίες που είναι πολύ περίπλοκες, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε κάποια κριτήρια ούτως ώστε να πετύχουμε μια βελτίωση. Επιπλέον θα πρέπει εμείς να υπογραμμίσουμε την αναγκαιότητα να σε αυτές τις δραστηριότητες να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτές που οδηγούν σε βιωσιμότητα και σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων. Από όλα θα πρέπει δηλαδή οι πιστώσεις για τις εξαγωγές θα, μπορέσουν, θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε επικροτώ την κατεύθυνση που ακολουθεί ο κύριος Σαντός στο έγγραφο εργασίας του. Νομίζω ότι είναι σωστή η κατεύθυνση αυτή. Διαφωνώ άρδιν με τον κύριο Κάσπαρη για τη γενική θέση του ΕΛΚ που θέλει να κάνει μια διάκριση ανθρώπινα δικαιώματα από τη διεξαγωγή εμπορικών δραστηριοτήτων. Όχι, δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Και όπως είπε και ο προλαλής σας, ο βαθμός της στήριξης των ποσών που δίνονται σε διεθνή κλίμακα είναι πραγματικά εκπληκτικός, προκαλεί δέος. Και φυσικά και έχει τεράστια επίπτωση σε πολλούς τομείς του κόσμου. Τα πρόσφατα γεγονότα, η καταστροφή παραδείγματος χάρη στον κόλπο του Μεξικού, θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο πιο προσεκτικά. Να δούμε μήπως θα έπρεπε να γίνει μια κριτική αξιολόγηση των έργων τα οποία δρομολογούνται, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα αποφευθούν στο μέλλον αντίστοιχες περιβαλλοντικές καταστροφές λόγω αυτών των εξαγωγικών πιστώσεων. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Ζαντό, ο αναφέρει το παράδειγμα του φράγματος Ελίζου στην Τουρκία που είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχει πτυχή ηθική, περιβαλλοντική, πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο αυτό το σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας του. Ίσως λοιπόν καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες για να ενδυναμώσουμε τις πτυχές αυτές, αλλά σίγουρα καλωσορίζουμε την κατεύθυνση που ακολουθεί Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα προσέξει τον Νικολό Ρινάλντι, συγγνώμη, που είναι σκιώδης εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα ιδιαίτερα πολιτικό το ζήτημα αυτό που θίγει έκθεση Ζαντό. Νομίζω ότι είναι λεπτό αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πραγματεύεται δε κάτι το οποίο μάλλον υπερβαίνει και το θέμα της ίδιας της έκθεσης. Γιατί το λέω αυτό. Το πρώτο πράγμα που με εκπλήσει είναι η διχοτόμια, η προφανής, που αναφέρει και το ίδιο το έγγραφο εργασία, αφενό μεταξύ νέα αρμοδιότητα, απληστική αρμοδιότητα ε, του Κοινοβουλίου για το εξωτερικό εμπόριο και αφετέρου μεταξύ τη διατήρησης και τις δράσεις, τις δράσεις ε, των ε, υπηρεσιών αυτών, ε, τις εξαγωγικές πιστώσεις. Είναι μια διχοτόμηση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει και θα πρέπει να υπάρξει σχετικός πολιτικός προβληματισμός στο πέσο της Επιτροπής μας. Και αυτός ο προβληματισμός υπερβαίνει τις κατευθυντήριες γραμμές. Δεύτερον, τα ποσά για τα οποία ε, πρόκειται για τις εξωτερικές αυτές πιστώσεις είναι τεράστια, είναι αστρονομικά ποσά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ασχολούμαστε με κάτι που αποτελεί πραγματικά κέντρα ε, οικονομικής εξουσίας, πυρήνες οικονομικής εξουσίας. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε από την άλλη. Η προσέγγιση του εισηγητή είναι σωστή. Επαναλαμβάνω όμως ότι Κατά την άποψή μου είναι κάτι που θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο των μελλοντικών μας δράσεων. Σε τρεις τομείς. Πρώτον, περίπλοκο νομίζω, ίσως προβληματικό, είναι το να υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα για το εξωτερικό εμπόριο από τη μια και από την άλλη να μην υπάρχει σχεδόν κανένα συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όλων αυτών των διαφορετικών οργανισμών. Δεύτερον, θα πρέπει να συμφωνήσουμε τουλάχιστον μεταξύ Ευρωπαίων στον ΩΣΑ για να δούμε ποια είναι τα κριτήρια εφαρμογής αυτών των ενισχύσεων για τις εξαγωγές. Το τουρκικό ζήτημα πράγματι αναφέρθηκε και στο έγγραφο εργασίας. Όταν μιλάμε όμως με τους διάφορους υπεύθυνους αυτών των ε, οργανισμών, Καθημερινά το βλέπουμε. Υπάρχουν δηλαδή οργανισμοί κάποιων κρατών μελών που λένε ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί υπερβαίνει τα κριτήρια που εμείς σεβόμαστε, περιβαλλοντικές ρήτρες κτλ. Και άλλα κράτη-μέλη, από την άλλη, θα τα χρηματοδοτήσουν τα έργα αυτά. Τρίτον, ενθαρρύνω τον εισηγητή και εδώ θα σταματήσω να ζητήσει να υπάρχει ως το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούς των υπηρεσιών αυτών. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο συντονισμού των δραστηριοτήτων μεταξύ των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων, γιατί εδώ μιλάμε για δημόσιο χρήμα. Αγγίζουμε μια κατάσταση αρκετά σκοτεινή από πλευράς διαφάνειας. Δεν υπάρχει λογοδοσία και αυτό πραγματικά είναι ανησυχητικό. κύριος Κάσπαρ έχει ζητήσει και πάλι το λόγο. Συνάδελφοι, να αναφερθώ σε κάποια από τα θέματα. Καταρχήν, παρακαλώ να γίνει η διάκριση ανάμεσα στην κατάσταση που επικρατεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει περισσότερη διαφάνεια από ό,τι σε άλλα όσον αφορά το μέσο αυτό, αλλά σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει και λιγότερη διαφάνεια. ό,τι και να θεσπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση και στα 27 κράτη-μέλη. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι το έγγραφο εργασία αυτό δεν ε, λαμβάνει υπόψη επαρκώ ε, την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεύτερον, το ΕΛΚ έχει ασχοληθεί με το θέμα των κοινωνικών προτύπων, των περιβαλλοντικών προτύπων κλπ. Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικά τα πρότυπα αυτά. Νομίζω όμως ότι επίσης συμφωνούμε ότι αν υπερβάλλουμε θα πετύχουμε ακριβώς το αντίθετο. Τι εννοώ. Αν έχουμε εξαγωγικές ε, πιστώσεις ε, για τομείς ε, όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις δικές μας που σέβονται τους ε, κανόνες μας, ε, τα ιδανικά μου, τότε ε, μπορεί αυτό τελικά να οδηγήσει στο αντίθετο. Και τέλος, το θέμα δεν είναι να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Γνωρίζω περίπου πώς εφαρμόζεται αυτό το μέσο στην Γερμανία. Θα πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε άλλα κράτη-μέλη. Βλέπω τον ε, συνάδελφο ε, Ρινάλη και άλλοι. Ε, δεν και ο πρόεδρος ζητά από τον ομιλητή να συντομεύσει. Μιλάμε για τι μικρομεσαίε που έχουν 15-20 συνεργάτε. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι το μέσο αυτό και όπως σας είπα πολύ ευχαρίστω στην κατάλληλη περίσταση θα ήθελα να συζητήσω το θέμα αυτό των εξαγωγικών πιστώσεων. Πιστεύω όμως ότι το συγκεκριμένο φάκελο δεν θα πρέπει να τον ε, φορτώσουμε με υπερβολικά πολλά ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας παρακαλώ να είσαστε όσο γίνεται σύντομος, διότι μας έχει τελειώσει ο χρόνος. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Τρία πράγματα έχω να πω αφού άκουσα τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα από πλευράς Επιτροπής, ως αρχή χαιρετίζουμε την έμφαση που η συγγετή σας δίνει στη διαφάνεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό που σχετίζεται με το εμπόριο. Δεύτερο σημείο, Φυσικά και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα εμείνουμε στην αρχική συλλογιστική γραμμή της πρότασής μας μεταφορά ε, των εθνικών ε, διατάξεων, στο, των κοινοτικών διατάξεων στο εθνικό δίκαιο. Θα δούμε ποιος είναι ο ανατολισμό του Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να είχαμε συνεργασία και με τα κράτη-μέλη και με το Κοινοβούλιο για πιθανή προσθήκη κάποιων διατάξεων. Κάποιες ε, τεχνικές διατάξεις θα είναι και εκτελεστές βέβαια, υποχρεωτικά και θα υπάρξει, ελπίζουμε, προστιθέμενη αξία στι απαιτήσει διαφάνεια που νομίζουμε ότι υπάρχει και σε ενωσιακό αλλά πολύ περισσότερο σε εθνικό επίπεδο. Τρίτον, Ελπίζουμε να μην υπάρξει ανισορροπία σε ό,τι αφορά τα προνόμια που μπορεί να έχουν τρίτες χώρες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας ε, τι τα συμφέροντα των εξαγωγέων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εισηγητής για τις τελευταίες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ε, έλαβα υπόψη όλα τα σχόλια. Εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει αυτό το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Είναι κάτι το καινούριο. Έχουμε τη συνομοθετική ιδιότητα το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες, για τις πιστώσεις ε, εξαγωγών και όπως και να έχει το θέμα, εμείς θα, προ... θα προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις σε σχέση με αυτό που μου ανησυχούμε, που μας ενδιαφέρει το θέμα της διαφάνειας και όπως είπαν ε, ε μερικοί σιώδες εισηγητές και είναι σημαντικό το θέμα, ε, το ότι χρειάζεται ένας έλεγχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μας επιβάλλει να μπορέσουμε να κοιτάξουμε, να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς γίνεται ακριβώς με αυτές τις υπηρεσίες. Τα ποσά, τα κονδύλια που επενδύονται είναι πολύ μεγάλα και γίνονται με βάση αξιολόγηση κινδύνων που είναι πολύ μεγάλη και γνωστή και υπογραμμίζω ξανά το θέμα της Αμερικής, ότι είμαστε πίσω σε σχέση με την Αμερική, με την αρμόδια Αμερικανική υπηρεσία. Ε, και θα πρέπει φυσικά να ε, κοιτάξουμε το ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν η συνεδρίαση. Το Σεπτέμβριο θα ξανασυζητήσουμε το σχέδιο έκθεση. Ολοκληρώνεται λοιπόν η δημόσια συνεδρίαση για σήμερα. Θα παρακαλέσω να παραμείνουν οι βουλευτέ ε, για τις συνεδρίες και κλεισμένων των θυρών και να εγκαταλείψουν την αίθουσα όλοι οι υπόλοιποι το συντομότερο δυνατό γιατί μα πιέζει ο χρόνο, παρακαλώ. Δηλαδή μόνο οι συντονιστέ θα παραμείνουν μαζί με τη γραμματεία, τη νομική υπηρεσία τους υπαλληλούς των πολιτικών ομάδων και η βοηθή των συντονιστών. Αυτοί μόνο μπορούν να παραμείνουν, όλοι οι άλλοι παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα. And also leave the discussions for the outside. Και ό,τι συζητήσεις έχετε παρακαλώ εκτός αιθούσης. This applies to the Commission also.